Liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Erstmal allen ein herzlich. Θα ήθελα να σας καλημερίσω όλους, να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας Τετάρτη απόγευμα που έχουν αρχίσει και φθήνουν σε μεγάλο βαθμό οι γραμμές εδώ στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας ε, σήμερα. Ειλικρινά δεν είναι καθόλου αυτονόητο και γνωρίζω ότι παραμονές ε, των διακοπών έχουμε πολλές υποχρεώσεις όλοι μας. Σας ευχαριστώ που ε, ήρθατε λοιπόν. Καταρχάς φυσικά θα ήθελα να πω ότι είναι η πρώτη πρώτη συνεδρίασή μας της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, πράγμα που σημαίνει ότι για ε, πρώτη φορά σήμερα θα ασχοληθούμε με την εξοικείωση ε, για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. Ε, έχουμε μεγάλο γλωσσικό καθεστώς σήμερα πολλές γλώσσες. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς και τους μεταφραστές για την εξαιρετική τους πάντα εργασία. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε προβλήματα ή διαφωνίες με την ημερήσια διάταξη, αν μπορούμε να προχωρήσουμε με το παρόν σχέδιο. Δεν διαφωνεί κανείς. Ωραία. Λοιπόν, δεύτερον, θέλω να καλωσορίσω θερμά τον Χέρνι Γκρέτεν που είναι μέλος του ε, ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, χαίρομαι που ξαναβλεπόμαστε, γνωριζόμαστε από παλιά. Ε, στη συνέχεια θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Λάζαρο Λαζάρου που είναι επίσης, δεν το βλέπω, α, εκεί πίσω δίπλα σας, από το ελεγκτικό συνέδριο και τον Μάρτιν Βέμπερ αριστερά σας, ε, διευθυντή των ελεκτρών. Α, ο κύριο Κρέτεν είναι στη μέση. Ωραία, πολύ ωραία, έχετε καθίσει. Θα σας δώσω μέσα στο λόγο, κύριε Κρέτεν για να μας κάνετε την πρώτη παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας πρόσκληση. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου του Προέδρου μα, Κλάου Χάινα Λένε, που δυστυχώ κολλείται σήμερα και δεν μπορεί να παρευρεθεί. Τον εκπροσωπώ εγώ, γιατί είμαι πρεσβύτερο εκεί στο ελεκτικό συνέδριο. Δεν θα χρειάζεται να με ανεχθείτε για πολύ ακόμα, γιατί στα τέλη του έτου λίγη η θητεία μου. Ε, με συνοδεύουν οι συνάδελφοι Λάζαρο Λαζάρου. Ο Λάζαρο είναι το αρμόδιο μέλος για την ετήσια έκθεσή μας. Εκείνον θα βλέπετε τους επόμενους μήνες πιο συχνά. Ε, και ο Μάρτιν Βέμπερ είναι ο διευθυντής ε, της Προεδρίας και θα τον ε, έχετε και εκείνο στην Επιτροπή σας και θα έχετε την ευκαιρία να το καλωσορίσετε ξανά. Σας ευχαριστώ και πάλι και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο τον Λάζαρο Λαζάρου για να σας ενημερώσει για την ετήσια έκθεση την οποία προβλέπουμε να εκδώσουμε στις 8 Οκτωβρίου και να σας την παρουσιάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνω μέσα στο λόγο ε, στον κύριο Λαζάρο, όπως είπατε κι εσείς. Thank you, Henri. Ευχαριστώ, Ανρή. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού, θα ξεκινήσω συγχαίροντάς σας όλους για την εκλογή ή επανεκλογή σας στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Και βεβαίω σα συγχαίρω εσάς όλο ιδιαίτερω πρόεδρε επειδή, ε, επί την εκλογή σας ε, ως πρόεδρο αυτή αυτής εδώ της Επιτροπής. Όπως είπε και ο συνάδελφο, είμαστε πολύ ευτυχείς που συμμετέχουμε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής σας. Συνεχίζουμε όπως ε, ανέκαθεν ε, τη συμβολή μας και την στήριξή μας στην άσκηση του ελεκτικού σας ρόλου. Θα με βλέπετε πολύ πιο συχνά από τον Οκτώβριο όταν μαζί με τον Πρόεδρο Λένε θα παρουσιάσουμε την ετήσια έκθεση. Εγώ είμαι μέλος υπεύθυνο για την ετήσια έκθεση και υπεύθυνο του πέμπτου τμήματος για τη χρηματοδότηση της Ένωσης. Κάνω αυτή την εργασία εδώ και τελευταία έξι χρόνια, οπότε θα έλεγα ότι είμαι ε, ήδη πολύ πεπειραμένο. Είχαμε πολύ αγαστή συνεργασία μέχρι τώρα και προσβλέπω στη συνέχιση της. Συντάσσουμε την ετήσια έκθεση, θα την υποβάλουμε στην Επιτροπή σας στις 8 Οκτωβρίου. Όπω ίσω ήδη να έχετε ενημερωθεί από τον Πρόεδρο Λένε, ε, τώρα είμαστε στην διαδικασία τροποποίησης της προσέγγισής μας όσον αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σταδιακά κινούμεθα προς ένα πρότυπο ε, βεβαίωσης όπου εκτός από την επιλογή των συναλλαγών και την παρακολούθηση των εμβασμάτων μέχρι το τελευταίο δικαιούχο ενθαρρύνουμε την Επιτροπή να προβεί σε κάποιες αλλαγές το σύστημα ελέγχου της, ώστε αν είναι όριμες ε, οι συνθήκες, εάν πληρώνται οι συνθήκες, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο την εργασία της Επιτροπής και των, και των ελεκτικών αρχών των κρατών μελών. Θέλουμε λοιπόν να δοκιμάσουμε ήδη και να ελέγξουμε τις εργασίες της Κομισιόν και των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών των κρατών μελών και να δούμε και ποια είναι τα αποτελέσματα των εργασιών που ήδη έχουν εκπονήσει αυτές οι εθνικές αρχές. Προβλέπουμε πως αυτή η προσέγγιση θα περικόψει τους πόρους που χρησιμοποιούμε για τον έλεγχο συμμόρφωσης, δηλαδή σε κάποιο στάδιο θα έχουμε περισσότερους πόρους ώστε να μπορούμε να κάνουμε πιο αποδοτική δουλειά. Επίσης, όπως τα γνωρίζετε, έχουμε ήδη αποφασίσει και από τον επόμενο χρόνο θα υποβάλουμε μια χωριστή ετήσια έκθεση σε σχέση με την απόδοση. Βέβαια, εγκαίρως πριν από τη διαδικασία απαλλαγής και Βεβαίως, με τα χαράς θα θέλαμε να έχουμε τη δική σας άποψη ε, όσον αφορά την απόδοση σε σχέση με τα σημεία που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Αυτό το project θα αναπτυχθεί με το χρόνο και ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε σε ένα στάδιο όπου θα δείτε προστιθέμενη αξία σε αυτήν την έκθεση. Τελειώνοντας λοιπόν θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε αυτή εδώ τη συνεδρίαση και θα ε, προσβλέπω ε, να σας δω και πάλι στις 8 Οκτωβρίου για την παρουσίαση της ετήσια μα έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πρώτα σας εισαγωγικά λόγια. Θα έχουμε πολύ εντατική συνεργασία από τον Οκτώβριο και μετά όταν θα κατατεθεί πλήρης έκθεση για το 2018. Χαίρομαι για τη συνεργασία που θα έχουμε και προσβλέπω σε αυτή. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μάρτιν Βέμπα. Παρακαλώ. Ε, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Χολμάγερ, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνάδελφοι της Γραμματείας Κοντ. Μετά τα εισαγωγικά λόγια των κυρίων Γκρέτεν και Λαζάρου, τώρα θα σας δώσω εγώ κάποια επιπλέον πληροφόρηση για το θεσμικό μας όργανο και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και την εργασία μας. Εδώ το πρώτο ζήτημα είναι πώς μπορούμε εμείς να σας βοηθήσουμε στη δουλειά που εσείς έχετε να επιτελέσετε. Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού παίζετε ένα ρόλο πρωταγωνιστικό 140 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως είναι τα ευρωπαϊκά χρήματα και θα πρέπει να φροντίζετε να, να ταπανώνται σωστά και με βάση κανόνες και προς το συμφέρον των 500 εκατομμύριων πολιτών. Εμείς, ως ελεγκτικό συνέδριο, έχουμε το ρόλο να σας βοηθήσουμε σε αυτό το πολύ δύσκολο έργο σας. Εμείς δεν είμαστε πολιτικό θεσμικό όργανο, αλλά τεχνικό. Δεν έχουμε εξουσία απόφαση ούτε μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις και ποινές για να τιμωρήσουμε εκείνου που δεν σέβονται τους κανόνες μας. Και σίγουρα δεν είμαστε και το πιο γνωστό ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Έχουμε όμως μια πάρα πολύ συγκεκριμένη εντολή ε, οικονομικού ελέγχου. Και ως εξωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δίνουμε ε, συμβουλές, διαβεβαιώσεις και αξιολογούμε τον κίνδυνο η εντολή μας ε, απορρέει από τις συνθήκες και μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε ανεξάρτητους ελέγχους σε όλα τα θεσμικά όργανα και τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο κρατών και περιφερειών και παγκοσμίω. Ε, οπουδήποτε δαπανώνται ευρωπαϊκά κονδύλια. Δηλαδή οι ελεγκτές μας πηγαίνουν όπου πηγαίνουν και τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανεξάρτητες ε, έρευνές μας με βάση στοιχεία δείχνουν ακριβώς τι συμβαίνει. Γι' αυτό παίζουμε ένα ε, ρόλο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο διαφανή και πιο λογοδοτούσα για να κατανοούν οι πολίτες τι συμβαίνει και που εκταμιεύονται τα χρήματα. Έτσι, βοηθούμε, πιστεύουμε, να διατηρείται η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο σημαντικό ίσως ε, σε ό,τι σας αφορά εσάς, τα ευρήματά μας, τα συμπεράσματά μας και οι συστάσεις μας μπορούν να σας βοηθήσουν εσάς, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως, να πάρετε τις εκάστοτε σωστές αποφάσεις για να αντιμετωπιστούν αδυναμίε και δυσκολίες που έχουν ανοιχνευτεί για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα οι πολιτικές και να προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί ε, παίζουμε ένα μοναδικό ρόλο στο θεσμικό πλαίσιο, γιατί η τεχνική μας δουλειά μπορεί να έχει πολιτικές συνέπειες. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή σας, Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, Προφανώ, εσείς είστε ο βασικό μα εταίρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικό μα σύμμαχος. Ε, οπότε συνεργαζόμαστε πολύ σκληρά και πολύ στενά. Έχουμε αφοσιωμένου υπαλλήλου που έχουν σχέσεις με το Κοινοβούλιο, είναι επιφορτισμένοι να είναι οι σύνδεσμοι, παρακολουθούν τις εργασίες τη επιτροπή σα ε, για να υπάρχει πολύ καλή ροή πληροφοριών και καλή ανταλλαγή ε, πάντα για να επικοινωνούμε εσείς και εμείς. Απευθύνω και ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους βουλευτές και της δικής σας Επιτροπής αλλά και άλλων. Πραγματικά μην διστάζετε να απευθύνεστε σε εμά όταν έχετε κάποιο θέμα που σας ενδιαφέρει. Υπάρχει ένα έθιμο μέχρι τώρα που δεν θα αλλάξει. Σε τακτά χρονικά διαστήματα ε, σας στέλνουμε ε, το χρονοδιάγραμμα για τις εκθέσεις που δημοσιεύουμε κάθε τρίμηνο και θα σας δίνουμε και πληροφορίες όσο χρειάζεται για την τρέχουσα εργασία. Θα στέλνουμε στην Πρόεδρο μια εμπιστευτική έκθεση, ένα αντίγραφο ε, και προς τους, ε, τη γραμματεία και τον εκάστοτε εισηγητή παραμονές της δημοσίευση της έκθεσης. Και άτυπα μπορούμε να συζητούμε με τους εισηγητές της εκθέσης μας πριν παρουσιαστούν εδώ στην Επιτροπή σας. Βεβαίω πάντα θα ερχόμαστε να παρουσιάζουμε και να συμβάλλουμε και σε ακροάσεις, συζητήσεις αλλά και διασκέψεις που διοργανώνεται εδώ και σε άλλες κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Θα ήθελα επίσης ε, σύντομα να σας δώσω επιπλέον πληροφορίες για κάποια σημαντικά στοιχεία της εργασίας μας στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πώς επιλέγουμε τα θέματα ε, για τον έλεγχο. Κάθε χρόνο επιλέγουμε κάποια θέματα με βάση την ανάλυση του κινδύνου που κάνουμε, λαμβάνοντας υπόψη ε, τα στοιχεία, τα αντικειμενικά ε, και το εκάστοτε ενδιαφέρον και στην αρχή του κάθε έτου απευθυνόμαστε στου εταίρου, καλούμε δηλαδή όλε τι επιτροπέ, τι κοινοβουλευτικέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μα προτείνουν ενδεχόμενα αντικείμενα για έλεγχο αυτό το αναλαμβάνει η διάσκεψη των πρόεδρων των επιτροπών, όπου τώρα προεδρεύει ο κύριο Σταγιάννη. Η δική σα επιτροπή συνεισέφερε πολύ σημαντικά ανέκαθεν ναι, σε αυτή τη διαδικασία και για φέτο, νομίζω, κάνατε γύρω στι 20 προτάσει για το πρόγραμμα εργασία μα για το 2020. Όπω ενημέρωσε ε, πέρυσι ο πρόεδρο Λένε, τον πρόεδρο τη επιτροπή ε, τη διάσκεψη των πρόεδρων των επιτροπών, το 40% των προτάσεων σας έχει καλυφθεί το 2019. Και περίπου το 60% της δουλειάς μας συνδέονται κάπως με προτάσεις και υποδείξεις και αιτήματα του Κοινοβουλίου προς εμάς. Αυτή τη στιγμή τώρα το ελεγκτικό συνέδριο εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας. Αυτό συμβαίνει συνήθως το φθινόπωρο κάθε χρόνο. Αυτό το χρονοδιάγραμμα ε, δημοσιεύεται και αποστέλλεται άμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως είπαμε και προηγουμένως, Έχουμε ένα τρίμηνο, ένα προγραμματισμό που αναφέρουμε πώς ε, πηγαίνει η, πρόεδρος, η πρόοδος των εργασιών συγγνώμη, και σας ενημερώνουμε και εσάς κυρία Πρόεδρε και τη Γραμματεία για να ε, κανονίσετε και εσείς το πρόγραμμά σας. Πώς αναφέρουμε λοιπόν τώρα ε, τα ευρήματα των ελέγχων που κάνουμε. Υπάρχουν διάφορες μορφές ελέγχων και αξιολόγησης καλύπτουν όλους τους ε, τίτλους του πολιτές δημοσιονομικού πλαισίου και όλους τους τομείς πολιτικής. Δηλαδή, έχουμε ελέγχου επιδόσεων για να δούμε ε, αν πιάνουν τόπο τα χρήματα. Ποιο είναι το παραγόμενο αποτέλεσμα σε σχέση με τους πόρους που διοχετεύονται εκεί. Συνήθως αυτές οι εκθέσεις φέρουν το τίτλο ειδικέ εκθέσεις. Επίσης κάνουμε και ελέγχους συμμόρφωσης και οικονομικούς ελέγχους στον προπολογισμό της Ένωσης και σε όλα τα θεσμικά όργανα οδηγούν αυτά σε δηλώσεις αξιοπιστίας ε, και εκεί εκφράζουμε ε, την άποψή μας για ε, ε, το κανονικό, το τυπικό, για τις πληρωμές, κατά πόσο υπάρχουν παρατυπίες, ατασταλίες κτλ. Καταθέτουμε μια δήλωση αξιοπιστίας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ετήσια έκθεσή μας. Αυτή η αλήθεια αξιοπιστίας και συμμόρφωσης όμως μπορούν να έχουν και τη μορφή ειδικών εκθέσεων. Εκεί συνεισφέρουμε στην ετήσια συζήτηση για την απαλλαγή που είναι η τελική έγκριση από το Κοινοβούλιο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μετά από τις συστάσεις του Συμβουλίου. Φέτος, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, η αιτήσια έκθεση θα έρθει να παρουσιαστεί στην Επιτροπή σας στις 8 Οκτωβρίου. Την τελευταία διετία έχουμε διευρύνει το εύρος των ε, προϊόντων που παρέχουμε για να αντιμετωπίσουμε διάφορες ανάγκες ενημέρωσης και έχουμε και αναλυτικά και περιγραφικά κείμενα για θέματα διαχείρισης. Έχουμε briefing papers ή διάφορες αναθεωρήσεις, επισκοπήσεις διαφόρων θεμάτων ή ειδικότερων θεμάτων ε, για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και τέλος, στις γνωμοδοτήσεις δίνουμε την άποψή μας για τη νέα νομοθεσία, για την αναθεωρημένη νομοθεσία, για νομοθετικές προτάσεις. Ε, ορισμένα αυτά εκδίδονται κατόπιν αιτήματος κάποιου θεσμικού οργάνου. Ε, όταν έχει αντίκτυπο στην οικονομική διαχείριση, αφορά τη συλλογή εσόδων, ε, αυτά είναι υποχρεωτικά και τα κάνουμε ιδία πρωτοβουλία. Πέρυσι, το 2018, Εκδώσαμε ρεκόρ δημοσιεύσεων εκτός από τις αιτήσεις εκθέσεις, 44 ειδικές εκθέσεις και αναθεωρήσεις και επισκοπήσεις και 10 γνωμοδοτήσεις. Ιδιαίτερα για τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έκτοτε έχουμε ε, κάνει ένα συμπίλημα ε, ε, σχόλια του ελεκτικού συνεδρίου ε, εν συντομία ε, λέγεται αυτό το έγγραφο και θα το βρείτε και στην ιστοσελίδα μας. Ε, πώς εξασφαλίζουμε την ακρίβεια των στοιχείων. Όταν μιλούμε για τον οικονομικό έλεγχο είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι πάντα διασταυρώνουμε τα στοιχεία και αυτά που αναφέρουμε είναι αντικειμενικά, είναι σωστά και όσο γίνεται ισορροπημένα και δίκαια. Συστηματικά έχουμε μία προσέγγιση που δεν εστιάζει στον ευνηδιασμό ε, και κατά την εκπόνηση των εκθέσεων. Δηλαδή, δίνουμε την ευκαιρία στον ελεγχόμενο ε, να σχολιάσει τα διάφορα στάδια του ελέγχου. Δεν υπάρχει νομική απέτηση να ε, καθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας και να τους διασταυρώσουμε μία φορά, αλλά εμείς το κάνουμε αυτό τουλάχιστον δύο φορές. Και όταν προβαίνουμε στις τελικές συστάσεις και συμπεράσματα, αυτά απορρέουν ε, από τις τελικές εκτιμήσεις και παρατηρήσεις και όχι από κάποιες δικές μας αρχικές εκτιμήσεις. Επιπλέον, στην ετήσια έκθεση και στις ειδικέ εκθέσεις ε, δημοσιεύουμε και τις απαντήσεις των ελεγχομένων. Αυτό δεν το κάνουν όλα τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια και οι εθνικές ελεκτικές αρχές. Και αυτό συνεισφέρει προς την αντικειμενικότητα και ισορροπία των εκθέσεών μας. Θέλω να πω και μερικά λόγια για το πολύ ευαίσθητο θέμα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφθορά θεωρείται μεγάλο πρόβλημα από πολλούς πολίτες για τον προπολογισμό και για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Το 2015, σε μια έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, περίπου 70% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι θεωρούσαν ότι ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υφίσταται ε, ε, συχνά ε, απάτες και το 60% απαντούσε ότι η διαφθορά ε, είναι σημαντικό πρόβλημα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Εμείς συνεργαζόμαστε πολύ ε, στενά με την Όλαφ, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Αντιμετώπισης Απάτης, παραπέμπουμε στην Όλαφ οποιαδήποτε ύποπτη περίπτωση για διαφθορά, απάτη, οποιαδήποτε άλλη παρανομία σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά το 2017, που ήταν το τελευταίο έτος που δημοσίευσαμε στοιχεία, ε, ε, δηλώσαμε στην Όλαφ 17 τέτοιες περιπτώσεις που είχαμε εντοπίσει. Και για το 2018 είναι αντίστοιχο περίπου το νούμερο. Εδώ είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι γενικά και μόνο για τη δήλωση αξιοπιστίας εξετάζουμε πάνω από 750 συναλλαγές. Ελέγχουμε. Δηλαδή, αυτό σας δείχνει και την τάξη μεγέθους. Ε, επιπλέον το τελευταίο 12 μήνο έχουμε εκδώσει τρεις εκθέσεις για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς. Μία για την Όλαφ και ε, την ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που δημιουργήθηκε πρόσφατα. Το δεύτερο στους ελέγχους κατά την πολέμηση απάτης ε, στα κράτη-μέλη για τη συνοχή και το τρίτο η καταπολέμηση του, της απάτης στο ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ποιες είναι οι στρατηγικές μας προτεραιότητες τώρα για το 2020. Το θεσμικό μας όργανο πρόσφατα γνώρισε πολλές αλλαγές τα τελευταία έτη. Και όλες αυτές οι αλλαγές έγιναν σύμφωνα με τις στρατηγικές προτεραιότητες που αποφάσισε το Κολέγιο των Ελεγκτών το 2017 για την περίοδο 2018-2020. Τώρα βρισκόμαστε στα μέσα της περίοδου. Όπως ακούσαμε προηγουμένως, κατά την τελευταία τριετία αρχίσαμε να αλλάζουμε την προσέγγιση μας για τη δήλωση αξιοπτησίας με βασική στόχευση να έχετε καλύτερη μέρωση για τη διαχείριση των οικονομικών και να είναι καλύτερη ιδίωση αξιοπιστίας. Μέσω μακροπρόθεσμα θα θέλαμε να προχωρήσουμε προς μία ε, διαδικασία πιστοποίηση σύμφωνα με τις διεθνείς ε, λογιστικές προ... προδιαγραφές ελέγχουμε και τα όσα μας λένε οι ελεγχόμενοι, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχέση με τις πληροφορίες που παίρνει και εκείνη από τα κράτη-μέλη, για παράδειγμα. Δύο χρόνια τώρα παρακολουθούμε αυτή τη νέα διαδικασία στα πλαίσια των ελέγχων της συνοχής. Ταυτόχρονα εστίαζαμε περισσότερο ε, στην αξιολόγηση των επιδόσεων της εκτέλεσης του προπολογισμού σε μια ευρία παλέτα, οικονομική και χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση, ασφάλεια και άμυνα και εξετάζουμε το μίσο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δρά ως ρυθμιστής κυρίως, όπως είναι η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα ή τα δικαιώματα των επιβατών, για να σας δώσω δύο παραδείγματα. Από τότε που εγκρίναμε τη στρατηγική μας για το 2018 μέχρι 2020, έχουμε κάνει και περισσότερους ελέγχους ε, επιδόσεων από ποτέ του χρόνου. Θα, ε, ε, από του χρόνου θα εκδίδουμε και μια ετήσια έκθεση ξεχωριστή για τις επιδόσεις. Επίσης, έχουμε αρχίσει κάποιε πρωτοβουλίε για να εντείνουμε τις ε, προσπάθειές μας προβολής, διαφήμισης ε, και ενημέρωσης του κοινού για να γνωρίζουν τα προϊόντα μας εδώ εισαγωγικών. Ε, διαφημίζουμε ακόμα περισσότερο τώρα τις εκθέσεις μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2018 παρουσιάσαμε 133 φορές διάφορα θέματα σε διάφορες επιτροπές, 65 στο Συμβούλιο και 15 σε Εθνικά Κοινοβούλια και μέχρι τώρα αυτό ήταν ο μεγαλύτερος αριθμό όλων των εποχών. Ταυτόχρονα έχουμε περισσότερες επαφές με τον τύπο και τα μίντια. Το 2018 μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων ε, βγάλαμε 76 δελτία τύπου και είχαμε γύρω στι 24 ενημερώσει τύπου. Επίσης επενδύσαμε πάρα πολύ στα social media και από ό,τι φαίνεται πιάσαν τόπο αυτές οι προσπάθειε Περίπου τριπλασιάστηκε η κάλυψή μας στα online media το 2018 και αναειδική έκθεση επίσης έχουμε μεγαλύτερη κάλυψη από τον τύπο από ό,τι στο παρελθόν. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι ε, εκδίδουμε περισσότερες εκθέσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες νομίζω έχετε αντίγραφα της έκθεσης πεπραγμένων μας για το 2018. Όπως όλες οι εκθέσεις μας υπάρχει και αυτή online και μπορείτε ανα πάσα στιγμή να εγγραφείτε στο newsletter, στο mailing list μας. Επίσης μπορεί και πάλι να σας φανεί χρήσιμο να κοιτάξετε το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ε, που σας δίνει μια ιδέα και μια γεύση για το τι προγραμματίζουμε και τι επίκειται για τους επόμενους μήνες. Συμπεραίνοντας, ελπίζω ότι κατάφερα να σας περιγράψω ορισμένα από τα στοιχεία της δουλειάς μας που να σας άνοιξαν την όρεξη να διαβάσετε τις εκθέσεις και να δείτε τη δουλειά μας έτσι λίγο πιο κοντά. Ελπίζω να πέρασα το μήνυμα ότι ο ρόλος μας ως Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο είναι μοναδικός, διότι η δουλειά μας μπορεί να είναι πολύ τεχνική, αλλά ε, μπορεί να έχει και πολιτικές συνέπειες. Αυτές οι συνέπειες φυσικά εξαρτώνται αποκλειστικά από εσάς που είστε εκλεγμένοι ε, εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών λαών. Εμείς μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε στη διάθεσή σας ε, για να Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά μετά τις στενές διακοπές για να βελτιωθεί η οικονομική διαχείριση και να ε, λειτουργεί καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος θα ήθελα να σας συγχαρώ και πάλι κυρία Χολμάια ξενόματος του Ελεκτικού Συνεδρίου και του Προέδρου Λένε που δυστυχώς σήμερα δεν μπορούσε να παρευρεθεί για την εκλογή σας ως ε, Πρόεδρος της Επιτροπής σας και την κυρία Μουνιώθ, την κυρία Κινίτσι ε, και τους επόμενους δύο αντιπρόεδρους ως αντιπρόεδρους και τον κύριο Ντότς. Και σας εύχομαι καλές διακοπές και ε, καλή επιτυχία στην κοινοβουλευτική περίοδο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. So, thank you very much. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική σας έκθεση και για ε, την ανάπτυξη του θέματος. Σας συγχαίρομαι και βεβαίως ε, ολόκληρη η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού αναμένει με ενδιαφέρον τη συνεργασία μαζί σας. Θα ρωτήσω τώρα τα μέλη μας, εάν ίσως κάποιος έχει ε, ερώτηση προς το ελεγκτικό συνέδριο. Ο κύριος Κούς. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και ε, το ελεγκτικό συνέδριο. Ερώτηση για την επιλογή των θεμάτων. Είπατε ότι δεν θα είναι η εργασία με χαρακτήρα πολιτικό. Όμως, από την άλλη μεριά, ομολογείτε ότι το έργο σας έχει πολιτικές επιπτώσεις. Πώς ε, αντιμετωπίζετε τον πειρασμό να επιλέξετε τα θέματα, ώστε επομένως να αποκτήσουν κάποια πολιτική απόχρωση. Ε, με την έννοια του ε, nudging, δηλαδή να μας ε, σπρώχνετε προς κάποια κατεύθυνση με την επιλογή των θεμάτων και τελικώς να καταλήξετε να είστε πολιτικός οργανισμός. Πώς το αποφεύγετε αυτό, η Πρόεδρος, η κυρία Βίντσικ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας και εκπρόσωπε του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είπατε ότι περνάτε από, την, από τον έλεγχο της συμμόρφωσης στον έλεγχο της επίδοσης. Επομένως, θα καθορίζονται στόχοι και θα ελέγχεται η επίτευξη του στόχου, για παράδειγμα έρασμος για νεαρούς επιχειρηματίες, αν δηλαδή φτάνει μέχρι περισσότερους επιχειρηματίες ή τι άλλο ακριβώ σημαίνει αυτό που μας εξηγήσατε. Τόμες, έχω την ίδια ερώτηση που είχαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοί μου, δηλαδή θα ήθελα να μάθω με ποιον τρόπο θα εγκρίνεται η επιλογή των στόχων και ποια θα είναι η μεθοδολογία των εκθέσεων. Γιατί θα συχνά για την αποτελεσματικότητα ε, των ευρωπαϊκών δαπανών και θέλω να μάθω πολύ καλύτερα με ποιον τρόπο από άποψη μεθοδολογίας θα συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα των ε, κονδυλίων, των δαπανωμένων κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Μαρτίνα, σας ευχαριστώ. Είμαι από τα παλαιότερα μέλη εδώ και θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο διότι πέντε χρόνια συνεργαστήκαμε με θαυμάσιο τρόπο και ε, συνιστώ στους νέους συναδέλφους και στις νέες συναδέλφους να συνεργαστούν στενά με το ελεγκτικό συνέδριο γιατί πάντοτε έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάσσουμε πληροφορίε κάνουμε και ετήσια κοινή συνεδρίαση. απλώ σύσταση εκ μέρου μου, γιατί πάντοτε μα φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμη η συνεργασία αυτή. Τώρα έχω δύο ερωτήσει. Στην προηγούμενη εντολή ε, καταβάλαμε προσπάθεια για την μείωση του χρόνου ε, των εκθέσεων, της ειδήσιας έκθεση και της έκθεσης MCA. Πώς μπορούμε τώρα να περάσουμε από το νη συν 2 στο νη συν 1 Γνωρίζουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι, αλλά πώ βλέπετε την δυνατότητα αυτή να συνεχιστεί η προσπάθεια και στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο να περιοριστεί, να χρονικά δηλαδή. Ήδη πετύχαμε πολλά, την συντομεύσαμε την περίοδο, αλλά όχι μόνο ένα μήνα. Πώ μπορούμε να κάνουμε περισσότερο, να γίνει ταχύτερη και να βελτιωθεί η συνεργασία και πολιτικά. Για το δεύτερο θέμα, πάντοτε εμένα με ενδιέφερε η performance η επίδοση των ε, ευρωπαϊκών δαπανών. Προτεραιότητα για μένα. Τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω ώστε να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ιδίως στις χώρες μέλη, διότι οργανώσαμε εργαστήρια, ακροάσεις, ε, ε, συνέδρια και από όλους τους φορείς και κυρίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έως τώρα, ωστόσο δεν έχουμε δει ουσιώδεις αλλαγές. Ε, βλέπουμε ευαισθητοποίηση, αλλά μπορείτε να προτείνετε και να κάνετε κάτι πιο συγκεκριμένο, ώστε να αλλάξει η επίδοση ε, της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Σας ευχαριστώ. Εσείς κύριε Βέμπερ τώρα. Να ανταποδώσω και εγώ τα συγχαρητήρια. Και ίσως να αρχίσω με το πιο απλό ερώτημα, πρώτο δηλαδή τη μεθοδολογία των ελέγχων μας. Και να πω μόνο ότι εάν σας ενδιαφέρει θα προσφέρουμε μια σειρά εργαστηρίων, θα προτείνουμε μια σειρά εργαστηρίων σε ε, κοινοβουλευτικού βοηθούς, συνεργάτες κλπ. για να εξηγήσουμε με περισσότερο λεπτομερή τρόπο πώς επιλέγουμε τα θέματα, πώς τα ελέγχουμε, πώς συντάσσουμε, συντάσσουμε τις εκθέσεις κλπ. Ε, να πω ακόμη ότι εργαζόμαστε ε, στην βάση γραπτών κατευθυντηρίων γραμμών που είναι και ε, διαθέσιμες εγγράφως στην ιστοσελίδα μας. Όποιος ενδιαφέρει ας τις αναζητήσει εκεί. Αλλιώς έλθετε σε επαφή μαζί μας ευθέω και ίσως θα μπορέσουμε να σας απαντήσουμε και ευκολότερα μάλιστα. Για το ερώτημα τώρα των performance audit, ίσως μπορεί να γίνει μετά μια συμπλήρωση από άλλους συναδέλφους μου, εγώ να έρθω αμέσως τώρα ερώτημα πώς να αποφευθεί δηλαδή ας πούμε μια πολιτική απόχρωση στα όσα πράττουμε. Πρώτα είναι σαφές ότι εργαζόμεθα μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο. Οτιδήποτε γίνεται εδώ άπτεται της πολιτικής. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολιτικό οικοδόμημα. Σε κάποιο βαθμό λοιπόν έχουμε και κάποια πολιτικά συμφραζόμενα. Όμως το έργο μας είναι κυρίως τεχνικό. Είναι αληθές βέβαια ότι επιλέγοντας κάποια συγκεκριμένα θέματα ρίχνει κανείς φως στα συγκεκριμένα αυτά θέματα αλλά ευαισθητοποιεί ε, το κοινό σε αυτά και ίσως όχι σε άλλα. Δεν μπορεί κανείς να καλύψει τα πάντα διότι και οι πόροι μας είναι περιορισμένοι. Όμως η διαδικασία προγραμματισμού μας είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να λειτουργήσει με τρόπο ισορροπημένο και ε, να είναι βασισμένη σε ενδείξεις, evidence-based, όσο είναι αυτό δυνατό. Δηλαδή έχουμε έναν μηχανισμό που μας επιτρέπει να αναλύουμε και να σταθμίζουμε τους διάφορους κινδύνους που βλέπουμε να αναφύονται σε διάφορους τομείς, να εξετάζουμε τις ε, οικονομικές επιπτώσεις των κινδύνων αυτών, δηλαδή αν κάτι πάει στραβά, ποιες θα είναι οι ζημιές, ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Και βεβαίως επιζητούμε να προστατεύσουμε τα συμφερόντα, τα συμφέροντα μάλλον των ε, ε, μετόχων μα εντό εισαγωγικών, δηλαδή Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων. Και λαμβάνουμε βέβαια και προτάσει και από εθνικά κοινοβούλια. Στη διαδικασία ε, για να καταλήξουμε στους περίπου 40 ελέγχου σε ένα έτος, προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε αυτές τις πτυχές. οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας έρχονται από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές μέσω των γραμματιών τους, απηχούνται όλες οι πολιτικές απόψεις, δεν απορρίπτουμε καμία πρόταση, διότι δεν ξέρουμε και από πού ε, προέρχονται ακριβώς, τις συλλέγει και τις προωθεί η διάσκεψη πρόεδρων ε, επιτροπών. Αυτό που κάνουμε είναι να ελέγξουμε εάν σηκώνουν έλεγχο, εάν είναι καθαρά πολιτικού χαρακτήρα η πρόταση σύσταση δεν θα της δώσουμε συνέχεια. Είμαστε ανεξάρτητος οργανισμός, τα μέλη μας προέρχονται και από τις 28 χώρες μέλη και αυτά λαμβάνουν τελικώς την απόφαση με τον πιο αντικειμενικό και ισορροπημένο δυνατό τρόπο. Η πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Εσείς τώρα κύριε Λαζάρου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις για τους ελέγχους επιδόσεων. Ας απαντήσω με μία σύντομη δήλωση, αν μου επιτρέπετε, γιατί θεωρώ ότι αυτή καλύπτει τα ειδικότερα ερωτήματα. Αυτό το performance auditing δεν είναι και τόσο εύκολος ο έλεγχος αυτός όπως ο οικονομικός έλεγχος ή έλεγχος συμμόρφωσης και δεν θα πρέπει να βάζουμε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή να εγείρουμε τις προσδοκίες πάρα πολύ ψηλά ήδη από τον πρώτο χρόνο, από το πρώτο έτος. Όπως εξήγησα προηγουμένως, θα συντάξουμε ετήσια έκδοση, έκθεση επιδόσεως για το 2019 το οικονομικό έτος 2019, αυτό θα γίνει επομένως σε ένα χρόνο από τώρα, ποσοτικοποιώντας δεν θα προσπαθήσουμε μάλλον να ποσοτικοποιήσουμε την επίδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο και εν πάση περιπτώσει με την διαδικασία πιστοποίησης που έχουμε ήδη ξεκινήσει attestation process ξεφεύγουμε από τον έλεγχο συμμόρφωσης. Η ετήσια έκθεση επιδόσεων, εκεί επιλέγεται μια εξελικτική προσέγγιση και συνεργαζόμαστε μαζί σας για να την βελτιώσουμε. Έως τώρα, ο AMPR, δηλαδή η ετήσια έκθεση διαχείρισης και επίδοσης που συντάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λόγω του χρόνου όπου τελικοποιήθηκε δεν μας επέτρεψε να την λάβουμε υπόψη στο ελεγκτικό μας έργο. Όμως από του χρόνου και επειδή η Performance Annual Report θα εκδίδεται λίγες εβδομάδες μετά από την ετήσια έκθεση, θα έχουμε τον χρόνο να επανεξετάσουμε τις πληροφορίες που θα μας έχει θέσει ε, στη διάθεσή μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τοποθετηθούμε. Άρα, ξεκινώντας θα παράσχουμε γνωμοδότηση προς εσάς για την αξιοπιστία και επάρκεια των πληροφοριών που θα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τα όσα κάνει και τα όσα ελέγχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, ε, υποτίθεται ότι έχει επιτύχει τους στόχους. Αυτά θα εξελιχθούν σύν χρόνο λαμβάνοντας υπόψη και την ανάδραση και το feedback που θα λαμβάνουμε από εσά. Εάν θεωρήσουμε ότι η ειδική έκθεση στοχευμένη στην επίδοση χρειάζεται περίπου 120 με 150 εβδομάδες ελέγχου εισέρχεται πλέον βαθιά στην επίδοση συγκεκριμένων τομέων πολιτικής. Και λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή πόρων για αυτή την ετήσια έκθεση επιδόσεων, που είναι δύο ή τρεις φορές μεγαλύτερη από τους πόρους που χρησιμοποιούμε για την ειδική έκθεση, για τις ειδικές εκθέσεις δηλαδή, δεν μπορεί να αναμένει κανείς τουλάχιστον στην αρχή, να προσφέρουμε μια ματιά πολύ σε βάθος για την επίδοση, για την επίδοση ενός ετήσιου προπολισμού της τάξης των 140 δισεκατομμύριων ευρώ. Επομένως, αρχικά θα είναι μια επισκόπηση στην βάση των πληροφοριών που θα παράσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σταδιακώς δε θα εξελιχθεί σε συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank. Gibt Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ε, σας ευχαριστώ. πρώτα, πρώτα, λοιπόν θερμά και με μεγάλη χαρά αναμένω την συνεργασία. Συμφωνώ άλλωστε απολύτω με αυτό που είπε η Μαρτίνα προηγουμένως ότι η συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο υπήρξε πάντοτε καρποφόρος και θετική. Ορίστε παρακαλώ, έχετε το λόγο και πάλι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο τελευταία λόγια. Όπως ήδη σας είπαμε, θα υποβάλουμε την ετήσια τη έκθεση στις 8 Οκτωβρίου. Ως ήθιστε, και εγώ ως ε, αρμόδιος για την ετήσια έκθεση, με χαρά θα συνεργαστώ πολύ πριν από αυτή την ημερομηνία με τον εισηγητή σας για την ετήσια έκθεση. Από ό,τι κατάλαβα, κυρία Πρόεδρε, θα είστε εσείς, η συγγήτρια, μάλιστα. Οπότε, από τα τέλη Αυγούστου, εγώ είμαι στη διάθεσή σας, μαζί με το επιτελείο μου, ώστε να συναντηθούμε και να σας ενημερώσω εκ των προτέρων για το τι θα περιέχει αυτή η ετήσια έκθεση, ώστε να είστε πιο καλά προετοιμασμένοι μόλις θα φτάσουμε στις 8 Οκτωβρίου και τις επόμενες συνεδριάσεις που θα ακολουθήσουν για τη διαδικασία απαλλαγή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος, για αυτή σας την προσφορά. Θα το εκμεταλλευτώ ώστε όντως να είμαι καλά προετοιμασμένη. για τα όσα θα μας απασχολήσουν τον Οκτώβριο. Σας ευχαριστώ και πάλι και προσβλέπουμε σε συνεργασία μαζί σας. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Αντέα Μπούσκι. Εσείς αντικαθιστάτε τον Διευθυντή. Έχετε ολόκληρη την ομάδα που γνωρίζω μέσω της Επιτροπής Προπολογισμού. Ε, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη αυτής της Επιτροπής, αγαπητά ε, τι ε, ε, μέλη του ελεκτικού συνεδρίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ για την εκλογή σας στο Ευρωκοινοβούλιο και σε αυτή την Επιτροπή όλος ιδιαίτερο. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου του κυρίου Κόπμαν, που είναι ο Γενικός Διευθυντής του Τμήματος για τον Προπολογισμό, αλλά δεν μπορούσε σήμερα να είναι εδώ. Η Επιτροπή αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί ελέγχει πολιτικά την εκτέλεση του προπολογισμού. Λογοδοτεί η Επιτροπή και η Κομισιόν το εκτιμά αυτό ιδιαίτερο. Είναι προ το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών και φορολογούμενων. Η διαδικασία απαλλαγή προσφέρει μια ευκαιρία για όλου του μετέχοντε να ε, προβληματιστούν για τι προηγούμενε ε, ε, για τις εξελίξεις, για τα γεγονότα, να δουν ποιε είναι οι καλύτερες πρακτικές και φυσικά να βελτιώσουν τη δημοσιονομική διαχείριση και να επιτύχουν καλύτερα από αποτελέσματα με τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Στη διάρκεια των ετών είδαμε θετικέ εξελίξει στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού, εκτέλεση μάλλον του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού, πράγμα το οποίο αντικοτοπτρίζει μια συνεχιζόμενη και επικοδομητική συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, τη δική σα Επιτροπή δηλαδή, το Συμβούλιο, την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Τα διδάγματα που αποκομίζουμε από το παρελθόν λαμβάνονται υπόψη στο σχέδιο ε, πρόταση για το επόμενο πολι πολιετές ε, σχέδιο. Ε, ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός εκτελείται από την Επιτροπή με κατόπιν προτάσεων των διαφόρων γενικών διευθύνσεων. Γι' αυτό και θα δείτε όλες αυτές τις, όλα τα τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ. Εντός της Επιτροπής ένας από τους βασικούς, τις βασικές ευθύνες της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού είναι να συνεργάζεται με την Επιτροπή ε, του Ελέγχου Προϋπολογισμού και την Επιτροπή προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και φυσικά και για να συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Η Επιτροπή ε, το τμήμα μας είναι υπεύθυνο, η γενική μας διεύθυνση είναι υπεύθυνη για το συντονισμό αυτής της συνεργασίας και ε, ε, με τα εξωτερικά όργανα, αλλά και εντός της Επιτροπής. Επιπλέον, η Γενική μας Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για τους δημοσιονομικούς κανόνες, για τον έλεγχο, τα ταμιακά, ε, τις δημοσιονομικές εκθέσεις και την προετοιμασία των ετήσιων λογαριασμών. Σήμερα είναι χαρά μου που, ακούω αυτό το τεχνικό, που, που συμμετέχω σε αυτό το τεχνικό εργαστήριο και βασικός μου στόχος είναι να σας δώσω μια γενική γενική εικόνα για τον προϋπολογισμό της Ένωσης από την έγκρισή του μέχρι την εφαρμογή του, την εκτέλεσή του και τον ελχό του. Η παρουσία σήμερα αρκετά εκτεταμένη, θα εστιάσω στα βασικά στοιχεία, αλλά πιστεύω πως είναι χρήσιμο για σας να δείτε αυτή την, την παρουσίαση PowerPoint, γιατί εκεί έχουμε πολλές πληροφορίες. Ο συνάδελφος θα ε, καλύψει ε, επίσης κάποια στοιχεία. Είμαι βεβαία ότι, έχουμε, ότι θα έχουμε επικοδομητικές σχέσεις στη διάρκεια της εντολής. Η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού είναι στη διάθεσή σας για να σας δώσει ε, πληροφορίες κάθε φορά που τις χρειάζεστε. Και μετά από αυτή την εισηγήση θα ήθελα να ξεκινήσω με την παρουσίαση PowerPoint. Όπως σας είπα, πρόκειται για έναν βασικό οδηγό ε, στον προπολογισμό του Ένωση. Θα ξεκινήσω με τα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Γιατί είναι τόσο διαφορετικός από τους προϋπολογισμούς ε, των ε, κρατών. Υπάρχουν τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του προπολογισμού. Το πρώτο είναι ότι είναι ένας επενδυτικός προπολογισμό. Δεν πληρώνουμε για υγειονομική περίθαλψη ούτε για συντάξει. Επενδύουμε μακροπρόθεσμα. Επίση, ο ευρωπαϊκό προπολογισμό φέρνει ε, προσθέμενη αξία συγκεντρώνοντα του πόρου του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα κράτη-μέλη μπορούν να επιτύχουν περισσότερα από ό,τι αν ενεργούσαν μόνα του το καθένα. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι ο ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι πάντοτε ισολογισμένο. Δεν μπορεί να υπάρχει προπολογισμό ο οποίο έχει έλλειμμα. Είναι ένα χαρακτηριστικό αδύνατο για τα κράτη-μέλη. Το συνολικό ποσό εσόδων είναι ταυτόσιμο με το, με το ποσό των πληρωμών. Τον... Και επίσης το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε έναν μακροπρόθεσμο προπολογισμό με βάση επταετίας. Αυτό που ονομάζουμε πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί έχουμε τόσο μεγάλο διάστημα, τι είναι το PDP, πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και γιατί χρειάζεται. Είναι η έκφραση των μακροπρόθεσμων πολιτικών προτεραιοτήτων. Δεδομένου ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, επενδυτικό για μακροπρόθεσμα και μακρόπνοα project, παρέχει με αυτόν τον τρόπο σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Και αυτό το κάνει όχι μόνο για τις δημοσιονομικές αρχές, αλλά και για τους δικαιούχους των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Έπειτα Πρόκειται για μια δέσμη που αποτελείται από τρεις πυλώνες. Ο πρώτο πυλώνας ο τρίτος πυλώνας είναι τα ποσά. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο κανονισμός περί ιδίων πόρων και το τρίτος πυλώνας είναι το νομοθετικό πρόγραμμα. Ο πρώτος πυλώνας είναι αυτός που είναι πιο γνωστός, ο πυλώνας των ποσών. Στο πολιετές ο βλέπουμε το σύνολο των εσόδων για το πολιετές πρόγραμμα και το μέγιστο ετήσιο ποσό που δύναται να δαπανίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια της περίοδου αυτής για κάθε κατηγορία δαπάνης. Αυτό ήδη προβλέπεται εξ αρχής για το PDP. Το PDP είναι δηλαδή το ανώτατο όριο. Δεν μπορούμε να δαπανήσουμε περισσότερα. Ο τρίτος πυλώνας είναι επίσης σημαντικός διότι αφορά το νομοθετικό πακέτο Μέσω του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου αποφασίζονται τα project και τα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και χρειάζεται γι' αυτό νομική βάση. Μέσα σε αυτή τη νομική βάση ε, επεξηγείται και ορίζεται ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιοι είναι οι στόχοι του κάθε project και όλες οι πληροφορίες που είναι σημαντικές για το κάθε πρόγραμμα. ενα 3 ευρώ είναι μεγάλος προπολογισμό δεν μπορεί να πει κανεί, αλλά στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει μόνο το 1% του συνόλου του ακαθάριστου εθνικού προϊόντο. και μόνο 2% των δημοσίων δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν συγκρίνουμε σε απόλυτα ποσά, για παράδειγμα για πέρυσι, είχαμε 150 δις είναι ένα ποσό χαμηλότερο από το συνολικό προπολογισμό του Βελγίου ή της Αυστρίας. Ακόμα και αν δεν είναι τόσο μεγάλος ο προπολογισμό, πετυχαίνουμε πολλά μέσω αυτού. Υπό το τρέχον ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή 2014 μέχρι 2020, έχουμε 187 δις για τις υποχρεώσεων και αυτό αυτά κατανέμονται με βάση τις πολιτικές προτεραιότητες. Το πρώτο ποσό είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και φυσική πόρη, δηλαδή βασικά γεωργία. Βλέπετε για πέρσι 39%. Το δεύτερο οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, 34%. Το τρίτο μεγαλύτερο ποσό είναι ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση, γύρω στο 13%. Ε, παγκόσμια Ευρώπη 6% η ασφάλεια και η θαγένεια και τέλος η διοίκηση. Πώς χρηματοδοτείται τώρα ο προπολογισμός. Ο προπολογισμός χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Έχουμε τριών ειδών ίδιους πόρους. Έχουμε τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους που είναι ε, κυρίως τελωνιακοί δασμοί που επιβάλλονται στις εισαγωγές ε, προϊόντων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ίδιους πόρους που από τον ε, φόρο προσθέμενης αξίας και τέλος έχουμε την ίδια σπόρους που βασίζονται στο ε, καθάριστο εθνικό προϊόν είναι το 1% και είναι το μεγαλύτερο ποσό το οποίο συμβάλλει στην ισορροπία ανάμεσα στα έσοδα και τις δαπάνες. Έχουμε επίση διορθωτικού μηχανισμούς που έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζουν τις υπερβολικά μεγάλες συμβολές από τα κράτη-μέλη. Ποιο ωφελείται, ποιοι είναι οι δικαιούχοι αυτών των ε, ε, ποσών αυτού του προπολογισμού. Έχουμε ένα σωρό δικαιούχου και εξαρτάται από τα διάφορα προγράμματα. Αλλά οι δικαιούχοι μα είναι εν γέννη ευρωπαϊκέ επιχειρήσεις, φοιτητέ και καθηγητέ, άνεργοι, επιστήμονες, περιφέρειες, πόλεις, γεωργοί, ΜΚΟ, τρίτες χώρες και όπως είπα έχουμε 6% ε, του προϋπολογισμού το οποίο απορροφάται από τις διοικητικές δαπάνες. Εδώ έχουμε μια γενική εικόνα του προϋπολογισμού και θα ήθελα επίσης να πω πώς εκτελείται ο προϋπολογισμός, γιατί τα ποσά είναι μεγάλα. Αν όλα εκτελούνται από την Κομισιόν, όχι. Το 1 τρίτο ε, εκτελείται από μάλλον, ε, συγγνώμη, ένα κομμάτι 20% εκτελείται από ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα κομμάτι κοινή διαχείριση, δηλαδή Κομισιόν και κράτη-μέλη, ε, δηλαδή είναι τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν μαζί, και το τελευταίο κομμάτι, έμεση διαχείριση από διεθνείς, οργανι... οργανισμούς και αποκεντρωμένους οργανισμούς, αλλά η Κομισιόν με την υποστήριξη των κρατών μελών είναι υπεύθυνη το σύνολο του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού και την εκτέλεση του. Γιώχαν τώρα θα σας εξηγήσει τον ετήσιο προπολογισμό. Ευχαριστώ, Ρώσα. Καλησπέρα σε όλους σας. Να σας δώσω μία επισκόπηση ε, για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώς έχει ενιάυσει η διαδικασία του προϋπολογισμού, πώς οργανώνεται και τι ε, ε, λέει σχετικά η συνθήκη, πώς ορίζει την όλη διαδικασία. Καταρχάς, δεν θα σας εκπλήξει που ο πυροπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εκτελείται στο κενό. Ε, είναι σαφές ε, και έχει οριστεί ξεκάθαρα στις συνθήκες τι μπορούμε να χρηματοδοτούμε και με ποιον τρόπο θα το χρηματοδοτούμε. Το ορίζει αυτό η συνθήκη η ίδια για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η συνθήκη ορίζει ακριβώς ποιε είναι οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να είναι αποκλειστικές ή συντρέχουσες αρμοδιότητες με τα κράτη-μέλη, αλλά αυτά ορίζονται σαφέστατα από τη συνθήκη και τι μπορεί ακριβώς να χρηματοδοτεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Από την άλλη βεβαίως υπάρχει ε, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο αιτία το PDP που καθορίζει το συνολικό μέγεθος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ε, οροφές ανατίτλο η κατηγορία και στον ίδιο τον κανονισμό αυτό εξηγεί και αναλύει σε ποιο βαθμό η ετήσια εκτέλεση μπορεί να αποκλίνει ε, από την αρμόδια αρχή, δηλαδή ποιος είναι ο βαθμός ευελιξίας. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το κανονισμό του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου που είναι ένα ογκώδε τεράστιο έγγραφο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί ανα που είναι πάντα αντικείμενο μακροσκελούς ε, ε, διαπραγμάτευσης ε, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου κατόπιν προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ορίζει πώς θα εκτελείται ο προϋπολογισμός σε λεπτομέρειες. Τι πρέπει να κάνουν οι φορείς για να εκτελέσουν τον προϋπολογισμό. Εδώ δεν αναφέρεται στη διαφάνεια, αλλά το είπε η Ρώσα προηγουμένως. η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού ορίζεται ε, μια απόφαση για τους ιδίου σπόρους. Και υπάρχει και οροφή στους ιδίου σπόρους που ξεπερνά το κανονισμό για το πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο. Διότι εκεί ορίζεται το απόλυτο ποσό δαπανών του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένου του PDP αλλά και των επιπλέον δαπανών αν θέλετε, αυτό είναι το ανώτατο όριο, το απότατο όριο, η οροφή. Next slide, please. Um, now who decides... Ποιος αποφασίζει λοιπόν σε αυτόν τον κύκλο του προϋπολογισμού. Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Με πολύ συγκεκριμένο τρόπο από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τρία διαφορετικά στοιχεία που καλύπτουν τρία διαφορετικά άρθρα της Συνθήκης. Σε ό,τι αφορά το μακροχρόνιο προϋπολογισμό, το μακροπρόθεσμο, έχουμε το άρθρο 312 που καλύπτει ε, τον κανονισμό, το δημοσιονομικό και ορίζει ότι ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να εγκρίνεται ομόφωνα από τα κράτη-μέλη αφού έχει ληφθεί η συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Article 312 το άρθρο 3.12. Μετά έχουμε την χρηματοδότηση του προπολογισμού, Είναι το άρθρο 3.11 της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει με ποιο τρόπο λαμβάνονται οι αποφάσεις για τους ιδίους πόρους. Και αυτό ε, συμβαίνει με ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών κατόπιν διαβουλεύσεως ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχουμε εδώ συνένεση, σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου, αλλά απλή διαβούλευση ratified by each. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να κυρώνονται όλα αυτά από κάθε κράτος ξεχωριστά σύμφωνα με τις συνταγματικές απαιτήσεις του κάθε κράτους. Δηλαδή η απόφαση για τους ιδίους πόρους συνήθως τίθεται σε ισχύ λίγα χρόνια μετά την επίτευξη συμφωνίας. Τρίτον, έχουμε την ετήσια ενιάυσια διαδικασία του προϋπολογισμού που ορίζεται στο άρθρο 314 της ΣΛΕ, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί βασικά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι ισότιμοι εταίροι στη διαδικασία λήψης της απόφασης, όπου το Συμβούλιο αποφάσει αποφασίζει με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία, δηλαδή δεν είναι ε, μομόφωνη αυτή η απόφαση. Και φυσικά το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την όλη διαδικασία και τον προπολογισμό. Και εκεί γίνεται και η τελευταία τυπική και επίσημη έγκριση του προπολογισμού. επανέρχομαι λίγο σύντομα στις λεπτομέρειες της ετήσιας διαδικασίας του προπολογισμού, άρθρο 3.14 της συνθήκης. Εδώ μιλάμε για το έτος νη πλην ένα. δηλαδή το έτος ε, πριν από τη χρονιά ε, του προπολογισμού. Αρχίζει με πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ονομάζεται σχέδιο Προπολογισμού και το οποίο κατατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα σχεδόν είτε κατά τη διάρκεια του μηνό Μαΐου είτε κατά τη διάρκεια του μηνό Ιουνίου. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει την πρότασή τη ε, μέσω των λεγόμενων τροποποιητικών επιστολών και κάθε χρόνο έχουμε τουλάχιστον μια τέτοια επιστολή η οποία ε, απευθύνεται, χρησιμοποιείται ε, για τη διόρθωση και την ενημέρωση των δαπανών για τη γεωργία. Αυτή η επιστολή έρχεται ε, συνήθως το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Μπορεί δηλαδή να τροποποιήσει μέχρι τέλειο Οκτωβρίου την πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η πρόταση λοιπόν, το σχέδιο προπολογισμού πηγαίνει πρώτα στο Συμβούλιο το οποίο τη συζητάει και εκφράζει άποψη. Εγκρίνει μια γνώμη και αυτή ονομάζεται η θέση του Συμβουλίου επί της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και στη συνέχεια, η ιστορία μας διδάσκει ότι συνήθως το Συμβούλιο περικόπτει την ε, πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παραδοσιακά. Και μετά τη στέλνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο με τη σειρά του ε, τροποποιεί την πρόταση του Συμβουλίου και πάλι η ιστορία μας διδάσκει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν δέχεται ποτέ τις περικοπές ε, όπως τις προτείνει το Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνήθως Ω πρώτο βήμα επαναφέρει τα αρχικά ποσά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και αναστέλει τι περικοπέ του Συμβουλίου και του ευγνωμονούμε πάρα πολύ εμεί ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά σύμφωνα με τι δικέ του προτεραιότητες βάζει και άλλε απαιτήσει με τροπολογίε για να ενισχυθούν κάποιοι τομεί και κάποιε δαπάνε. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν προτείνει πάντα αυξήσεις. Καμιά φορά το Κοινοβούλιο μπορεί να προτείνει και περικοπές. Το έχει κάνει ήδη. Το παράδειγμα που είναι πολύ πρόσφατο και έχω υπόψη μου ήταν πέρσι όταν πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημαντική περικοπή της προενταξιακής βοήθειας ε, για την Τουρκία. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιστρέφει στη συνέχεια στο Συμβούλιο και πάλι διδασκόμαστε από την ιστορία ότι το Συμβούλιο δεν τα δέχεται αυτά, τα απορρίπτει και απορρίπτοντας την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτόματα μπαίνουμε στη φάση της λεγόμενης συνδιαλλαγή. Εκεί συναντώνται τα τρία θεσμικά όργανα, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθούν να βρουν μια συμφωνία για τον προπολογισμό. Okay. There was a, small hiccup here. Έπαθε ένα λόξι το μηχάνημα εδώ. Here. The Φέτος η συνδιαλλαγή προβλέπεται από τις 29 Οκτωβρίου μέχρι τις 18 Νοεμβρίου. Και η πρόεδρός σας έχει πολλή δουλειά μπροστά της, διότι δεν είναι απλώς αρμόδια για τον προϋπολογισμό του 2018, αλλά είναι και γενική εισηγήτρια του προϋπολογισμού για το 2020. Άρα θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Καμιά φορά αποτυγχάνει και η συνδιαλλαγή σε μερικέ χρόνια. Οπότε αναγκάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει τέλη Νοεμβρίου ένα νέο σχέδιο προϋπολογισμού και εκεί έχουμε μια υπερταχεία διαδικασία για να ε, προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε. Μετά δε τη συμφωνία αυτή, ο προϋπολογισμός ψηφίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγκρίνεται και υπογράφεται από τον πρόεδρό του κανονικά στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. Δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες και ποσά ε, του προπολογισμού για το 2019. Ίσως να πούμε μόνο ότι για τον προπολογισμό του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 1,5% ε, αύξηση στην ανάληψη υποχρεώσεων. Το Συμβούλιο περιέκοψε 1,5 δισεκατομμύριο και το Κοινοβούλιο θα γνωμοδοτήσει μετά το καλοκαίρι από αυτού. Αφού εγκριθεί ο ετήσιος ευρωπαϊκό προπολογισμό πρέπει να και να εκτελεστεί. Άρα είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι στη διάρκεια της εφαρμογής του προϋπολογισμού της εκτέλεσης γίνεται σωστή διαχείριση, αυτή είναι η επιτυχή της συμμόρφωσης και το δεύτερο τμήμα είναι ότι, επιτυχάνουμε ότι θα πρέπει να επαληθεύσουμε και να ελέγξουμε ποια είναι τα αποτελέσματα επιτόπου και ποια είναι η επίδραση και οι επιπτώσεις στους πολίτες. Απόδοση δηλαδή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και αυτό έχει να κάνει με την ερώτηση που τέθηκε πριν από λίγο. Ποια είναι τι είναι ο προπολογισμό απόδοση, τι είναι το πλαίσιο απόδοση. Η έννοια δεν είναι τόσο περίπλοκη. Η έννοια αυτή είναι να έχουμε ένα πλαίσιο ότι για κάθε πρόγραμμα θα έχουμε ένα σύνολο στόχων, ένα σύνολο προτεραιοτήτων και <clears throat> κάποια μέσα με τα οποία να εκτιμούμε και να αξιολογούμε αν οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν. Ποια είναι ε, όμως τα μέσα που έχουμε στη διαθέσή μας να ελέγξουμε την επίτευξη των στόχων είναι διάφοροι δείκτες απόδοσης και επίσης κάνουμε διάμεσες αξιολογήσεις στα μέσα δηλαδή τα, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Με όλες αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να αξιολογήσουμε αν προχωρούμε στη σωστή κατεύθυνση, αν ε, ε, εκτελείται σωστά ο προπολογισμό και αν επιτυχάνουμε ε, τους στόχους που, έχουν αποφασίσει, που έχει αποφασίσει ο νομοθέτης. Η ιδέα δεν είναι δύσκολη, αλλά η εφαρμογή ε, ε, του προπολογισμού απόδοσης ε, έχει, μέσα, περιέχει πολλές προκλήσεις. Πρώτη πρόκληση είναι ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Για χρόνια όλοι εστιάζαμε στο κομμάτι της συμμόρφωσης. Θέλουμε ε, τώρα να συνεχίσουμε το, με το τμήμα αυτό της συμμόρφωσης, αλλά να εστιάσουμε και περισσότερο στο ε, κομμάτι της απόδοσης. Και αυτό είναι αλλαγή νοοτροπίας όχι μόνο στο επίπεδο της Επιτροπής, στο επίπεδο και των διεγούχων και των κρατών μελών. Και δεύτερον, θα πρέπει να εντοπίσουμε στόχους και δείκτες σχετικούς. Είναι εύκολο, αλλά κάποιες φορές δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο να εντοπίσουμε ευφυείς δείκτες που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, ε, σωστά για την αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, να εντοπίσουμε δε δείκτες όπου να έχουμε τις πληροφορίες. Ο προπολογισμό μα εκτελείται σε 28 κράτη-μέλη αλλά και εκτός Ένωσης ε, και πρέπει εμείς να μπορούμε να συλλέγουμε όλες τις πληροφορίες που προέρχονται από όλους τους δικαιούχου. Είναι μεγάλη πρόκληση για μας και τα κρατημέλη, αλλά και για όλα ε, τις τους ε, συμμετέχοντες, όλους αυτούς τους φορείς που σας ανέφερα για να μπορούμε να σας ετοιμάσουμε και τις εκθέσεις μας γιατί ο απότερος στόχος είναι να έχουμε στη διάθεσή μας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να λάβουμε αποφάσεις μέσα στην διάρκεια του πολιετούς και για το επόμενο πολιετές. Η πολιετής φύση του προπολογισμού είναι και μια από τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακριβώς επειδή αρχίζουμε την εφαρμογή του προπολογισμού ένα χρόνο αλλά θα φαντάζεστε ότι τα αποτελέσματα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα διαθέσιμα. Ξεκινάμε τον πρώτο χρόνο, εκτελούμε τα προγράμματα που είναι διετή ή τριετή και τα πρώτα αποτελέσματα θα τα έχουμε σε τρία χρόνια. Πραγματικός αντίκτυπος δηλαδή θα ε, φανεί πολύ αργότερα. Και αυτή είναι μια από τις ιδιαιτερότητες του προϋπολογισμού, ότι δηλαδή... σκεφτόμαστε σε αιτήσια βάση, αλλά ο προπολογισμό είναι πολυετή. Αυτή η πτυχή πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όχι μόνο από εμά, αλλά και από εσά, όταν θα συζητάμε κάθε φορά μέσα στο πλαίσιο τη διαδικασία απαλλαγή. Μέσα στο τρέχον πολιετέ έχουμε περίπου 250 στόχους και 700 δείκτε. Πιστεύουμε πως είναι υπερβολικά πολλοί. Αυτό το σύστησε και το Ευρωκοινοβούλιο και το Ελεκτικό Συνέδριο, πως θα ήταν καλύτερο να περιοριστεί ο αριθμός των στόχων και ο αριθμός των δικτών. Και αυτή η σύσταση ελήφθη υπόψη για το επόμενο πολιετές. Έχουμε μειώσει πολύ τον αριθμό των στόχων και έχουμε προσπαθήσει να εντοπίσουμε τους καλύτερους δείκτες. Υποθέτω ότι αυτό, αυτή την πρόταση της Κομισιόν θα την στηρίξετε, γιατί στόχος θα είναι, στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης για την νομική βάση, κάθε θεσμός θα ήθελε να προσθέσει και άλλους στόχους και άλλους δείκτες. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα προσκρούσουμε στο ίδιο πρόβλημα που έχουμε και τώρα στο τρέχον. PDP. Η Κομισιόν λοιπόν καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το τομέα της απόδοσης για τις εκθέσεις και την επικοινωνία ε, είναι ε, ένας από τους τομείς που έχουμε προχωρήσει πολύ. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι βασικά υπάρχουν δύο ειδών έγγραφα τα οποία αφορούν την απόδοση. Το πρώτο είναι το πρόγραμμα και ε, είναι μάλλον οι προγραμματικές δηλώσεις που δημοσιεύονται μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού και όπου εξηγώνται όλες οι ιδιαιτερότητες του πλαισίου απόδοσης για κάθε πρόγραμμα τα, ε, οι προγραμματικές οι προβλέψεις αυτές ε, οι προγραμματικές ε, είναι αυτές όπου περιγράφεται η κατάσταση απόδοσης κάθε προγράμματος. Πρόκειται για ένα έγγραφο που δείχνει ποιες είναι οι επιδόσεις στη διάρκεια του τρέχοντος PDP και είναι και αυτό κάτι που συμβάλλει στη διαδικασία απαλλαγής. Τώρα θα ήθελα να στραφώ σε μια άλλη έκθεση που είναι πολύ σημαντική γιατί όλες οι εκθέσεις ε, και η λογοδεσία είναι σημαντικά για την Ένωση. Μιλήσαμε λοιπόν για την απόδοση αλλά έχουμε και την πτυχή τη δημοσιονομική. Ετησίως υιοθετούμε τους αιτήσιους λογαριασμούς είναι αυτή που μπορεί να βρει κανείς σε μια ιδιωτική εταιρεία ή σε εταιρείε ε, του δημόσιου τομέα. Οι αιτήσιοι λογαριασμοί ε, ε, προετοιμάζονται από το λογιστικό μας τμήμα και υιοθετούνται κάθε χρόνο από την Κομισιόν και επίσης αυτή έχουμε εκεί ισολόγιο, έχουμε το παθητικό, το ενεργητικό, αυτή, ο αιτήσιος αυτός λογαριασμός ελέγχεται από εξωτερικό ελεγχτή και από το ελεγκτικό συνέδριο. Τα τελευταία 11 χρόνια έχουμε λάβει γνωμοδότηση ε, καθαρή, ας το πω έτσι, για τους ετήσιους μας λογαριασμούς. Εξηγούμε πώς δουλεύουμε λοιπόν για την απόδοση, ότι είναι πολύ σημαντική και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη όλες τις συστάσεις που έχουμε λάβει από το Κοινοβούλιο και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά έχουμε και το, το κομμάτι της συμμόρφωσης που για πολλά χρόνια δουλέψαμε πολύ σε αυτό. Όπως είπα, η Κομισιόν είναι ο ίστατος υπεύθυνο για την εκτέλεση του προπολογισμού. Ακόμα και αν αυτό γίνεται σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, Όπω είπα, ο προπολογισμό εκτελείται με διάφορα, σε διάφορα τμήματα, αλλά η Κομισιόν πρέπει να αναλαμβάνει ευθύνη και είναι εκείνη που λογοδοτεί για την εκτέλεση του προπολογισμού. Πώς είμαστε σε θέση λοιπόν να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Αυτό γίνεται τη βάση επί τη βάση ενός ε, μοντέλου διαχείρισης. Έχουμε όμως και τους δικούς μας αρμόδιους ε, ελεγκτές, το εσωτερικό μας έλεγχο, ε, έχουμε τους εσωτερικούς διατάκτες και έχουμε και τους ελεγκτές του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και έτσι εξασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση. Εδώ αυτό το, το σχήμα που βλέπετε φαίνεται περίπλοκο, αλλά δεν είναι στην ουσία, γιατί αποτελείται από τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι το επιχειρησιακό ε, σκέλος, της Ο δεύτερος πυλώνας είναι η ε, λογοδοσία του Κομισιόν και έχουμε και ένα τρίτο πυλώνα εξωτερικό που είναι ο εξωτερικός έλεγχος του προπολογισμού που ασκείται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και το πολιτικός έλεγχος που ασκείται από το Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα, το πρότυπο ε, αξιοπιστίας είναι διαφορετικό από αυτό που εκδίδει το ελεγκτικό συνέδριο γιατί εμείς το βασίζουμε από, σε ένα σύστημα που λειτουργεί από κάτω προς τα πάνω. Έχουμε ένα σωρό ελέγχους ε, που μας δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να ε, τροφοδοτήσουμε αυτά τα τμήματα που συναποτελούν την αξιοπιστία. Κάθε Γενικός Διευθυντής ε, ετοιμάζει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, όπου βρίσκουμε πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς έχει εκτελεστεί ο προπολογισμό από κάθε γενική διεύθυνση. Κάθε γενική διεύθυνση επίσης πρέπει να πει εάν υπάρχουν αδυναμίες και ποιες είναι οι δράσεις που θα ήθελε να εφαρμόσει ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος για το κομμάτι της συμμόρφωσης. Με όλες αυτές τις πληροφορίες έχουμε το διατάκτη, έχουμε το γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου και τότε η Κομισιόν ε, ε, ε, εγκρίνει την ετήσια έκθεση διαχείρισης όπου έχουμε και απόδοσης. Έχουμε δύο κομμάτια, ένα για την συμμόρφωση και ένα για την απόδοση. Μετά την έγκριση αυτού, ε, τότε η Κομισιόν αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Επίσης, οι Επιτροποί, εγκρίνουν ε, μία δέσμη για πρώτη φορά στο Δημοσιονομικό Κανονισμό. Έχουμε το ολοκληρωμένο, την ολοκληρωμένη δέσμη λογοδοσίας. Πρόκειται για ένα σύνολο πληροφοριών που στόχο έχουν τη διαδικασία απαλλαγής. Εδώ θα βρείτε μόνο πληροφορίες που χρειάζεστε για να δείτε πώς έχει εκτελεστεί ο προπολογισμό στο πλαίσιο του PDP. Τώρα, όπως σας είπα, ε, το σύστημά μας ξεκινά από κάτω προς τα πάνω. Εδώ έχετε ένα παράδειγμα που αφορά την γεωργία. Έχουμε λοιπόν αυτά όλα τα στοιχεία ώστε να φτιάξουμε το αξιοπιστία. Έχουμε πρώτον τις, ε, ε, τους οργανισμούς πιστοποίησης, μετά έχουμε τις, τους οργανισμούς πληρωμών, το σώματα ε, πιστοποίησης και μετά έχουμε την Κομισιόν. Έχουμε και πρέπει να ελέγξουμε τα είδη δαπανών, έχουμε διάφορα προληπτικά αλλά και διορθωτικά μέτρα. Ε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών. Τα προληπτικά μέτρα είναι αυτά που, γίνονται, που, που εφαρμόζονται πριν να εκτελεστούν, πριν να γίνουν ε, τα εμβάσματα κτλ. Και τα διορθωτικά μέτρα είναι αυτά που γίνονται αφού έχουν καταβληθεί οι πληρωμές, γιατί είναι αδύνατον εκ των προτέρων να ελέγξουμε τα πάντα. Υπάρχουν δηλαδή εκ των προτέρων έλεγχοι και εκ των υστέρων έλεγχοι. Στα προληπτικά μέτρα εντάσσονται οδηγίες, εκπαίδευση, ε, κατάρτιση, αλλά και διακοπή και αναστολή των πληρωμών, αν βρούμε πολλές αδυναμίες. Στα διορθωτικά μέτρα έχουμε, εφόσον εντοπίσουμε αδυναμίες και ανακτούμε τα χρήματα μέσω ε, ε, διαταγών ανάκτησης. Ο στόχο είναι να προστατεύσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και υπάρχει μηδενική ανοχή για απάτη. Σφάλμα δεν σημαίνει απάτη. Σφάλμα μπορεί να σημαίνει ότι κάποιες πτυχέ, ας πούμε, σε, μια, σε ένα δημόσιο διαγωνισμό, κάποια στοιχεία να μην είναι απόλυτα σωστά. Το ποσοστό όμως σφάλματος δεν είναι τόσο μεγάλο. Έχουμε έναν απότατο στόχο στην εφαρμογή, στην εκτέλεση του προπολογισμού. Ο απότατο στόχο είναι στο τέλο των προγραμμάτων, όταν όλα τα προγράμματα πια έχουν ολοκληρωθεί και κλείσει, ο τελικός κίνδυνος αντικανονικότητα αντικανονικότητας όσον αφορά τη συμμόρφωση είναι κάτω του 2% γιατί είναι το, αυτό το ανώτατο κατόφλι που επιτρέπει το ελεγκτικό συνέδριο. Αυτή η αξιοπιστία που θέλουμε να έχουμε με στόχο κάτω του 2% είναι σημαντικό εκεί να λάβουμε υπόψη τον πολιτή χαρακτήρα εκτέλεση του προπολογισμού, διότι όπως είπα τα προγράμματα διαρκούν πολλά χρόνια, κάνουμε πληρωμές για το ίδιο πρόγραμμα και το ίδιο project σε διάρκεια 2, 3, 4 ετών και οι έλεγχοι δεν γίνονται όλοι πριν καταβληθούν οι πληρωμές. Έχουμε έλεγχο ε, και μετά την καταβολή των ποσών. Και γι' αυτό τον λόγο μπορεί να υπάρξουν σφάλματα ή κίνδυνοι. Τη στιγμή των πληρωμών ή τη στιγμή του ολοκλήρωσης. Αλλά για μας είναι πιο σημαντικό το τέλος. Γιατί στο τέλος του προγράμματος κάθε φορά είναι σημαντικό ο κίνδυνος αντικανονικότητας να είναι χαμηλότερος από το 2%. Όπως σας είπα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να λειτουργεί εν πλήρη διαφανεία. Και όταν διάφοροι διατάκτες ε, εντοφίζουν σημαντικές αδυναμίες στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, κάθε ένας διατάκτης θα πρέπει να το αναφέρει αυτό και να κάνει κάποιες παρατηρήσεις και όλες αυτές να τις αποκαλύπτει στην ε, ετήσια έκθεση πεπραγμένων και όλα αυτά ε, περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες εκθέσεις και επιδόσεων. Είναι ένας τρόπος να ενημερώνονται και οι πολίτες και η δημοσιονομική αρχή όταν έχουν εντοπιστεί σοβαρές αδυναμίες. Λογοδοσία και διαφάνεια διέπει όλη τη δράση μας και συνοψίζεται σε αυτή. Είναι σημαντικό αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να λογοδοτούμε, είμαστε υπόλογοι και θέλουμε να είμαστε και διαφανείς. Και κάθε χρόνο εγκρίνει ε, μια ε, ε, δέσμη μέτρων, ένα πακέτο το οποίο εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2018 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπήκε για πρώτη φορά πέρσι στο δημοσιονομικό κανονισμό και μέσα στη δέσμη αυτή, αυτό το πακέτο, έχουμε πέντε βασικές εκθέσεις. Η πρώτη είναι η αιτήσια έκθεση διαχείρισης και επιδόσεων. Εξηγήσαμε και τις επιδόσεις και τις, τη διαχείριση. Έχουμε τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Επίσης, Έχουμε την αιτήσια ε, ε, έκθεση για τους εσωτερικούς ελέγχους, μια έκθεση που είναι σημαντική για το Κοινοβούλιο, η συνέχεια που δίνεται στη διαδικασία απαλλαγής του προηγουμένου οικονομικού έτους γιατί το Κοινοβούλιο χορηγεί την απαλλαγή ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αυτή συνοδεύεται και από ένα ψήφισμα με διάφορες συστάσεις, τις οποίες υλοποιεί όλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης έχουμε μία έκθεση για τις μελλοντικέ εισρωές και εκροές. Ε, τι προβλέπουμε μέσα στην επόμενη πενταετία να γίνει. Έτσι, μια πρόβλεψη είναι, μια προβολή ε, για το πώς θα εκτελεί το προπολογισμό μέσα σε μια πενταετία. Με αυτή τη δέσμη λοιπόν το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο αλλά και οι πολίτες έχουν όλες τις προφορίες για το πώς εκτελέστηκε ο προπολογισμό κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Και αυτή η ε, δέσμη εκθέσεων που θα παρουσιάσει το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, ο Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό, ο κύριος Έτιγκερ, είναι σημαντική για τη διαδικασία ε, της απαλλαγής. Έτσι αρχίζει η διαδικασία της απαλλαγής. Παρουσιάζει αυτό το πακέτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ελεκτικό Συνέδριο μάλλον ε, την ετήσια έκθεση, γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων ε, επιτρόπων και κοινοβουλίου και έχουμε και όλες τις συστάσεις του Συμβουλίου. Όλα αυτά είναι στοιχεία που σειραίουν στη διαδικασία της απαλλαγής και βοηθούν το Κοινοβούλιο να τη χορηγήσει. Μέχρι εδώ όλα αυτά είναι εξήγηση της τρέχουσας κατάστασης ε, και του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Πριν ολοκληρώσω όμως έχει σημασία, κυρίως για τα νέα μέλη, να δώσουμε λίγο μια ενημέρωση για το τι συμβαίνει με το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα σας τα πει αυτά ο Γιώχαν Ουρέλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για την περιγραφή των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την διαδικασία. Και θα παραμείνω στην επιφάνεια γιατί είναι περίπλοκο το θέμα με πολλές συνιστώσεις. Τον προηγούμενο Μάιο εγκρίναμε πακέτο με διάφορα στοιχεία, κυρίως τις εξής συνιστώσεις. Πρόταση νέου κανονισμού MFF, δεύτερο πρόταση για νέα διαθεσμική συμφωνία, τρίτο πρόταση για νέα απόφαση για ιδίους πόρους. Αυτές είναι οι βασικές συνιστώσεις της δέσμης που πρόκειται να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συμφωνίας. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η πρότασή της είναι και φιλόδοξη αλλά και ρεαλιστική. Και βεβαίως εκλήθημε να λάβουμε υπόψη ότι κάνουμε μια πρόταση για μια Ευρώπη των 27 και όχι των 28 πια. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της Βρετανικής αποχώρησης και του κενού χρηματοδότησης που θα αφήσει πίσω της αυτή η αποχώρηση. Η Κομισιόν έκανε πρόταση η οποία ανταποκρίνεται σε 1,11% του ΑΕΠ των χωρών μελών, μαζί και με την πρόταση εγγραφή στον προπολογισμό των όσων βρίσκονται εκτός, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αναπτύξεως. Αυτό το 1,11% κρίθηκε υπερβολικά γενναιόδωρο από το Συμβούλιο Υπουργών και βέβαια ανεπαρκές από το Κοινοβούλιο. Η μάλλον όπως εξήγησε προηγουμένως η Ρώσα για το πλαίσιο επιδόσεων, performance framework, που είναι επίσης μια σημαντική συνιστόσα των προτάσεών μας και ιδίω λόγω του περιορισμένου μεγέθους του κοινοτικού προϋπολογισμού έχει σημασία να στοχεύουμε επενδυτικά στους τομείς εκείνους όπου υπάρχει δυνατότητα να προσφερθεί προσθέμενη αξία. Κάναμε προσπάθεια επίσης να απλοποιήσουμε τους κανόνες να τους κάνουμε πιο συνεκτικούς και γενικά να μειώσουμε την γραφειοκρατική επιβάρυνση εις βάρος των δικαιούχων. Και τέλος, στις προτάσεις μας περιλαμβάνουμε και ορισμένα πρόσθετα μέτρα, τα οποία θα συμβάλλουν σε μεγαλύτερη ευκαμψία και μέσα στα ίδια τα προγράμματα, αλλά και μεταξύ τους. Και ενισχύουμε και τα εργαλεία για την αντιμετώπιση ε, κρίσεων και ε, απροβλέπτων. Στην πρότασή μας περιλαμβάνουμε μια νέα δομή με 7 τίτλους που ε, συμβαδίζουν και με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Δεν θα σας τα πω όλα τώρα με λεπτομέρεια, αλλά αυτό που έχει σημασία, κατά τη γνώμη μου, είναι να σημειώσει κανείς ότι μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, απλούστευσης προσπαθήσαμε να μειώσουμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, δηλαδή ε, των τομεακών νομοθεσιών, από 58 σε 37. 58 σε 37. Πρόκειται για σημαντική μείωση. Ορισμένα από τα πιο σημαντικά νέα στοιχεία της προτάσεώς μας και δεν θα πω βέβαια σε λεπτομέρειες ούτε και εδώ σας τα αναφέρω μόνο για να τα γνωρίσετε είναι η πρόταση να ιδρυθεί ο μηχανισμός Invest EU, Invest EU που θα είναι ένα οριζόντιο ταμείο που θα περιλαμβάνει όλα τα ε, υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, πολύ σημαντική νέα πρόταση, καθώς και την πρόταση να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο. Στο τομέα των εξωτερικών προτείνουμε ένα ε, συνολικό οριζόντιο μηχανισμό που να συνεργαστεί και με τους μηχανισμούς γειτονίας κλπ. και να περιλάβει όλα τα εφιστάμενα εργαλεία για δράσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, με εξαίρεση την προενταξιακή βοήθεια. Για τους μηχανισμούς διαχείρισης συνόρων και μετανάστευσης θα έχετε ακούσει περισσότερη την πρόταση που άλλωστε έχει εγκριθεί από Κοινοβούλιο και Συμβούλιο για τη δημιουργία μιας ε, διαρκούς ε, δύναμης 10.000 συνοριοφυλάκων, καθώς και ε, ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή, ευρωπαϊκή δηλαδή ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή. Σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την ευκαμψία δηλαδή, είναι προτείνουμε ένα κοινοτικό αποθεματικό, νέο δηλαδή εργαλείο ευκαμψίας που μαζί με τα υφιστάμενα μας επιτρέπει να ανακυκλώνουμε ε, αποδεσμευμένα κονδύλια από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό ήταν διαρκής απέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει περιληφθεί λοιπόν στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του προπολογισμού, την απόφαση για τους ιδίους πόρους, έχουμε λάβει υπόψη ε, τις ε, ανέκαθεν απαιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προτείνοντας έναν αριθμό νέων ιδίων πόρων, που έχει μεγάλη σημασία νομίζω αυτό για το Ευρωκοινοβούλιο και δεύτερο, από τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, συγγνώμη, που το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει σύντομα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που αποκαλούμε ε, η μητέρα όλων των επιστροφών, δηλαδή η Βρετανική επιστροφή θα πάψει να υπάρχει και θα συμπαρασύρει και τις άλλες υφιστάμενες επιστροφές. Βλέπετε στην στη διαφάνεια που προβάλλομαι τώρα, <clears throat> βρίσκω ότι έχει ενδιαφέρον γιατί δείχνει από τη μεριά του πρώτου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου υπό τον ε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Delors το 1988 βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο έχει κινηθεί έχουν κινηθεί δαπάνες πάνω-πάνω βλέπετε την σημασία της κοινή αγροτικής πολιτικής να μειώνεται, θα έλεγα σχεδόν ε, διαρκώς σταδιακά. Η μεσαία καμπύλη είναι οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, η οποία αυξήθηκε πολύ σημαντικά ε, στο πρώτο και δεύτερο ε, πολιετή δημοσιονομικά πλαίσια, μετά λίγο πολύ έγινε οριζόντια και τώρα κάπως αρχίζει να μειώνεται. Και αυτό βέβαια απηχείται και στη σημαντική αύξηση της βαρύτητας των άλλων προγράμμων, εκεί, ε, προγραμμάτων. Εκεί βλέπετε other programs. Και υπό την ισχύ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, αυτά τα τρία θα έχουν την ίδια βαρύτητα. Στον προϋπολογισμό η δε τελευταία καμπύλη είναι μάλλον σταθερή και ε, αντιπροσωπεύει την διοικητική δαπάνη. Να μην σας στερήσω επίσης μια σύντομη επισκόπηση των θέσεων του Κοινοβουλίου για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο του Κοινοβούλιο. Στις 18 Νοεμβρίου ενέκρινε προσωρινή έκθεση όπου προτείνει το επόμενο πι να αυξηθεί σε 1,3% του ΑΕΠ δηλαδή 16-17% παραπάνω από αυτό προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ορισμένα από τα ε, πιο σημαντικά στοιχεία προτεραιότητας στην έκθεση αυτή του Κοινοβουλίου είναι πρώτο κοινή αγροτική πολιτική και συνοχή να διατηρηθούν σε πραγματικούς αριθμούς και αντίθετα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου σε πραγματικούς αριθμούς και λαμβάνοντας υπόψη και το βάρος του πληθωρισμού προβλέπεται μείωση για αυτές τις δύο αρκετά παραδοσιακές πολιτικές. Το Κοινοβούλιο επίση προτείνει σημαντική ενίσχυση για το ορίζον Ευρώπη και το έρασμος ΣΥΝ και πέραν δηλαδή των ενισχύσεων που προέβλεπε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σημαντικό επίσης για το Ευρωκοινοβούλιο είναι ότι ε, επιθυμεί πιο φιλόδοξους στόχους για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, δηλαδή για τι σχετικέ δαπάνες στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και μάλιστα με τον καιρό που κάνει τώρα έξω, μου φαίνεται αρκετά ορθή αυτή η απέτηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει επίσης και στον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ενδιάμεσης αναθεώρησης. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνδέει την συνενεσή του για τον κανονισμό πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου την συνδέει δηλαδή με την εισαγωγή νέων πόρων. Έρχομαι σιγά σιγά στο τέλος της παρουσιάσεως και θα σας δώσω μια πολύ σύντομη επισκόπηση για το πού βρισκόμαστε. Η διαφάνεια σας δείχνει πού βρίσκονται οι ε, διαπραγματεύσεις για τις νομικές βάσεις ανατομέα. Θα δείτε στο πράσινο 12 προτάσεις που έχουν κατά βάση φτάσει σε μερική συμφωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων των δύο συνομοθετών δηλαδή, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Αναμένουμε την συμφωνία για το ΠΔΠ να τελικοποιηθεί δηλαδή. Ο, ο ορίζον Ευρώπη είναι επίση πολύ σημαντικό μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η διασύνδεση της Ευρώπης σε κίτρινο χρώμα οι προτάσεις όπου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο είναι έτοιμα να αρχίσουν τους τριμερείς διαλόγους και σε πορτοκαλί και ερυθρό, εκεί τα πράγματα έχουν προχωρήσει λιγότερο. Απόλυτα τελευταία διαφάνεια είναι το χρονοδιάγραμμα, όπου βρισκόμαστε τώρα υπό φιλανδική προεδρία, από την πλευρά δηλαδή του ε, Συμβουλίου. Οι επερχόμενες προεδρίες βασίζουν τις εργασίες τους ε, σε αυτό που λέγεται ε, πλαίσιο διαπραγματεύσεων, negotiating box, που τον Οκτώβριο θα καταλήξει στην δημοσίευση εγγράφου που θα περιλαμβάνει αριθμό σημείων που θα συζητήσουν σε βάθος τα δύο θεσμικά όργανα τον Οκτώβριο με την ελπίδα η συμφωνία να υπάρξει μεταξύ των μελών του Συμβουλίου πριν από το τέλος του έτους. Και φτάνουμε τότε πλέον στην άνοιξη του επομένου έτους για την συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό την ε, διαδικασία σύμφωνης γνώμης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή που χαρίσατε στα λόγια μου. Η Ρόζα. Η παρουσίαση σας δείχνει ότι ο προπολογισμό αναφέρεται και στο παρελθόν και στο παρόν και στο μέλλον. Τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε με τη διαδικασία απαλλαγή 2018, εκτελούμε το προπολογισμό του 2019 και συζητούμε το επόμενο ΠΔΠ 2021 2027. Θα ήθελα να πω ότι η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να συνεχίσει η επικοδομητική συνεργασία με την Επιτροπή σας. Σας προσφέρουμε επίσης, αγαπητή κυρία Πρόεδρε και βεβαίω και σε όλα τα μέλη σας, εάν χρειάζεστε άλλες πληροφορίες, εάν θεωρείτε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε με άλλο τρόπο, είμαστε στη διάθεσή σας ανά αντικείμενο. Έχουμε ετοιμάσει και ένα πακέτο για όλα τα μέλη της Επιτροπής σας με όλες τις πληροφορίες για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό σε περισσότερε λεπτομέρειε από ό,τι ήταν δυνατό να εξηγήσουμε σήμερα. Το επόμενο βήμα μας θα είναι η παρουσίαση από τον Επίτροπό μας κύριο Έτινγκερ τον Σεπτέμβριο για το πακέτο περί λογοδοσίας που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλωστε βρισκόμαστε εδώ ενώπιόν σας και για να απαντήσουμε και σε άλλες ερωτήσεις εάν έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα και εσάς, ε, κύριε Μποσχέτσα, αλλά και τον κύριο Ουρέλ, ε, τον οποίο συνεργάζομαι ε, ανέκαθεν πάρα πολύ στενά. Και σας ευχαριστώ για την τόσο ζωντανή παρουσίαση και την τόσο περιστατωμένη και ακριβή. Ερωτήσεις έχουν οι συνάδελφοι. Ε, ο κύριος Σαστέλ. Στα γαλλικά θα μιλήσω, μα φυσικά, λίμωνο. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους διάφορους ε, ομιλητές από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι γεγονός ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος του προϋπολογισμού είναι βασική λειτουργία για να έχουμε καλύτερη διαχείριση των ε, δημοσίων οικονομικών και τη βέλτιστη ακριβώς διαχείριση των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων και μια καλή θεσμική, διαθεσμική συνεργασία. Ασία πραγματικά θα ε, πρέπει να βελτιώνει την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την αποτελεσματικότητα. Πόσο μάλλον που η Ευρωπαϊκή Ένωση ζει κρίσιμε στιγμές. Βλέπουμε και από το Brexit ότι στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει δύσκολες επιλογές. Ε, και θέλω να επιμείνω το εξή. Γενικά, οι Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις εκθέσεις που μας διαβιβάζουν εστιάζουν στα σημαντικότερα και τα πιο ενδιαφέροντα για την Επιτροπή μας για να διευκολύνουν την εργασία μας. Το ίδιο ισχύει και επιμένω για να έχουμε τις ίδιες προτεραιότητες κατά την ακρόαση των διαφόρων γενικών διευθυντών της Επιτροπής. Η κυρία Βίντσικ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Στα αγγλικά να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Νομίζω ότι είπατε ότι ο υπολογισμό ε, είναι 150 δισεκατομμύρια ετησίως, αντίστοιχο με τον αυστριακό προπολογισμό. Ω πρώην πρόεδρος ε, της Επιτροπής Προπολογισμού στη Βουλή μας, πρέπει να ε, είμαι ειλικρινή, είναι μόλις 80 δισεκατομμύρια ο προπολογισμό τη Αυστρίας, όχι 150. Άλλε ερωτήσει έχετε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τότε να ξαναδώσω το λόγο ξανά στην κυρία Μπουσκέτση και στον κύριο Ουρέλ. Πρώτον για την αποτελεσματικότητα των εκθέσεων και τα σημαντικά και μετά για τα νούμερα. Ευχαριστώ για αυτό το σχόλιο για τον προϋπολογισμό της Αυστρίας. Βλέπω ότι στη διαφάνεια αναφέρεται διαφορετικό ποσό ε, είναι από μια επίσημη ιστοσελίδα, αλλά θα το διασταυρώσουμε και θα το διορθώσουμε. ναι, αφού έχουμε αυστριακούς συναδέλφους, εντάξει, το είχαμε βάλει εντός εισαγωγικών, εντός παρενθέσεων. Σε ό,τι αφορά το σχόλιο του κυρίου Ολιβιέ Σαστέλ, Απαντώ στα γαλλικά. Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάρα πολλές πληροφορίες. Όπως σας είπα, είναι πέντε οι εκθέσεις ε, σε αυτή τη δέσμη λογοδοσίας και διαφάνειας. Νομίζω ότι θα είχε σημασία επίσης και για μας να γνωρίζουμε ε, ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες και τα σημαντικότερα σημεία. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε και εμείς να συνεργαστούμε με τους γενικούς διευθυντές και τους διαφόρους επιτρόπους όταν έρχονται εδώ στις διάφορες ακροάσεις ακριβώς για να εστιάσουμε στα θέματα που εσείς θεωρείτε σημαντικότερα. Εμείς μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιες προτεραιότητες και αυτά που εμείς θεωρούμε σημαντικά. Καλό θα ήταν όμως εκ των προτέρων να τα συζητούμε μαζί σας για να έχουμε ε, τη βέλτιστη δυνατή ε, συνεργασία. Πριν έρθουν για τις ακροάσεις λοιπόν οι γενικοί διευθυντές και οι επίτροποι, καλό θα ήταν να το δούμε λίγο διμερώς, ε, ποια είναι τα θέματα που σας ενδιαφέρουν εσάς περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Νομίζω ότι η ιδέα του κυρίου Σαστέλα έχει πολύ μεγάλο νόημα. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε ε, εμεί τα μέλη της Επιτροπής μας, τις προτεραιότητές μας, τα σημαντικά θέματα που θα μας απασχολήσουν και τα βασικά ζητήματα. Και θα τα διευκρινίσουμε μετά και σε συνεννόηση μαζί σας. Θα σας πούμε ποιες είναι οι σημαντικότερες προτεραιότητες για τους βουλευτές. Βεβαίως είναι αυτό εκ των όνων για να είναι καλύτερη και πιο επιτυχημένη η συνεργασία μας και η δουλειά μας εδώ. Άλλες ερωτήσεις έχετε? Όχι. Να προχωρήσουμε λοιπόν. Αφού ακούσαμε το ελεγκτικό συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτενώς, έχουμε και άλλη δυνατότητα οι βουλευτές εμείς να ενημερωνόμαστε, να αναθέτουμε μελέτες και λοιπά και έρευνες και αυτό είναι οι δικές μας υπηρεσίες. Έχουμε την επιστημονική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, την οποία είχα την ευκαιρία να χρησιμοποιήσω επανειλημμένα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Νίλς Φίσερ για την παρουσία του εδώ μαζί με το επιτελείο του και να δώσω μέσω το λόγο αλλά προηγουμένως θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τη Βέρα Μιλισέβιτς και τον Ρούρο Φαρσαρτίνς, πυρογνώμονες για τις επιτροπές, τον Ρον Κόρβερ από το EPRS για τη ε, ε, μονάδα, το τμήμα ε, ελέγχο εκ των υστέρων για τις εκθέσεις εφαρμογών και τον Αλισάντο Νταλφόνσο, EPRS, ε, θέματα δημοσιονομικά και πραγματογνωμοσύνη ε, και εμπειρογνωμοσύνη μετά από αίτημα των μεμονωμένων βουλευτών. Ο κύριος Φίσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που έχουμε να έρθουμε να σας ενημερώσουμε τόσο νωρίς στην κοινοβουλευτική περίοδο, ιδιαίτερα τα νέα μέλη, ε, να σας ε, παρουσιάσουμε τις διάφορες δυνατότητες που έχουμε και θα το γυρίσω τώρα στα αγγλικά. Να σας δώσω τώρα μια σύντομη ε, εισήγηση για τον τρόπο με τον οποίο ζητούμε και λαμβάνουμε εμπειρογνωμοσύνη τόσο από τους εμπειρογνώμονες εντός του Ευρωκοινοβουλίου όσο και και από αυτούς εκτός. Όπου μπορούμε να αναθέσουμε εξωτερικές μελέτες και ε, ενημερώσεις. Δεύτερη διαφάνεια παρακαλώ. Υπάρχει, μια βασική, υπάρχει ένας βασικός διαχωρισμός για το πώς μπορούμε να ζητήσουμε εμπειρογνωμοσύνη. Έχουμε δηλαδή δύο τρόπους. Από τη, στα ε, αριστερά βλέπετε τα κοινοβουλευτικά όργανα όπου έχουμε τα ε, τμήματα πολιτικής όπου παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη στις, προς τις επιτροπές και άλλα κοινοβουλευτικά ε, όργανα. Να σας αναφέρω εν συντομία γιατί είναι έτσι οργανωμένα. Όταν εγώ εργάζομαι ως βοηθός κάποιο ευρωβουλευτή, εργαζόμουν ως βοηθός ευρωβουλευτή πριν από πολλά χρόνια, ο ευρωβουλευτής μου είχε μια σπουδαία ιδέα για μελέτη για την Επιτροπή δηλαδή ε, προπολογισμού. Ε, κάλεσε τότε την ε, υπηρεσία και τότε εκείνη η υπηρεσία του είπε ναι, σπουδαία ιδέα, αλλά είναι Νοέμβριος. Εμείς είμαστε ήδη πλήρεις. Έχουμε το πρόγραμμα εργασίας για το επόμενο χρόνο. Αν θέλετε, το μεθεπόμενο χρόνο θα ανταποκριθούμε στην πρότασή σας. Όπως ε, γνωρίζετε, τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου δεν θέλουν να περιμένουν δύο χρόνια, όπως φαντάζεστε μάλλον, δεν θέλουν να περιμένουν δύο χρόνια πριν να ε, ε, έχουν αυτές τις εμπειρογνωμοσύνες που θέλουν, τις μελέτες που θέλουν. Τώρα όμως συνδέεται η, το αίτημα για μελέτη με τη συνεχιζόμενη εργασία, την εξε, υποεξέλιξη εργασία νομοθετική και κοινοβουλευτική επιτροπή. Στα δεξιά βλέπετε το δεύτερο τρόπο για να ζητήσει κανείς κάποια μελέτη είναι για μεμονωμένα μέλη. Εάν δηλαδή έχετε ένα αίτημα για μια συγκεκριμένη έρευνα, που όμως δεν συνδέεται άμεσα με κάποιο επίκαιρο θέμα, ε, δεν θέλετε να ζητήσετε από τον συντονιστή, μπορείτε να το κάνετε με αυτόν τον τρόπο και να ε, ρωτήσετε από την υπηρεσία ερεύνης των Ευρωβουλευτών. Να σας παρουσιάσω τώρα σύντομα τους συναδέλφους που θα σας ε, ενημερώσουν πιο συγκεκριμένα για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ζητάτε κάποια μελέτη έρευνα. Εδώ στα δεξιά μου Βλέπετε τον κύριο Μάγκη, που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Συνεχίζουμε Εδώ βλέπετε τη τέταρτη διεύθυνση, τη, τη, διεύθυνση ΔΕΛΤΑ για ε, τα δημοσιονομικά θέματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι όντως τα τμήματα ε, πολιτικής συνεργάζονται στενά με τα κοινοβουλευτικά όργανα, δηλαδή επιτροπές και τις διευθύνσεις που εργάζονται ε, για νομοθετικούς και άλλους φακέλους. Η ΕΞΠΟ είναι διαφορετικά οργανωμένοι. Έχουν ένα τμήμα πολιτικής που καλύπτει όλες τις επιτροπές και αντιπροσωπείες. Ενώ στις εσωτερικές πολιτικές είναι διαρρεμένο σε πέντε. Και στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε ότι μέσα στη Διεύθυνση Δημοσιονομικών Υποθέσεων έχουμε τρεις μονάδες και όντως πρόκειται περί στενής συνεργασίας. Κάτι που είναι ενδιαφέρον να σημειώσει κανείς είναι ότι όντως κάποιες φορές στο τμήμα πολιτικής έχουμε μια κάπως καλύτερη εικόνα των επιτροπών ε, ε, προπολογισμού και ελέγχου προπολογισμού από ότι κάθε μία ξεχωριστά γιατί τείνουν να εστιάζονται στη δική τους ε, εργασία. Προχωρώ. ποια είναι η αποστολή του Τμήματος Πολιτικής. Να δίνει έγκαιρη και ειδικευμένη ε, ενημέρωσης και συμβουλές σε επίκαιρα θέματα. Είμαστε στη διάθεση των επιτροπών από τη στιγμή που οι συντονιστές ζητήσουν κάποια μελέτη ή μπορεί να είναι και ο πρόεδρος. Ε, η αντίδρασή μας είναι άμεση. Εάν γίνεται εξωτερική έρευνα, ε, παίρνει κάποιο περισσότερο χρόνο γιατί δεσμευόμαστε από τον δημοσιονομικό κανονισμό τον οποίο ξέρουμε πάρα πολύ καλά και που διευκρινίζει πώς γίνεται το καθετί. Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες συμβάσεις για τις ε, που προβλέπονται από τις διαδικασίες και τα μεγαλύτερα project παίρνουν περισσότερο χρόνο τόσο όσον αφορά τη διαδικασία όσον αφορά και τους ερευνητές ε, ή τους μελετητές που είναι εξωτερικοί. Και Είμαστε ένα think tank, όπως είναι και το EPRS. Είμαστε μικρότερο, αλλά ε, ε, είμαστε πιο κοντά στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Εδώ έχουμε λοιπόν κατά παραγγελία υπηρεσίες, όπως τις ε, βλέπετε, κάθε μία μελέτη πρέπει να έχει εγκριθεί από τους συντονιστές. Εμείς διαχειριζόμαστε το οικονομικό κομμάτι Και αυτό μπορεί να αφορά ενημέρωση και μελέτε όχι μόνο για τις επιτροπές αλλά και τον πρόεδρο, τις των επιτροπών, τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα. Έχουμε οριζόντια συνεργασία και project, έχουμε δηλαδή επαφή με τους ε, διάφορους ε, θεσμούς. Ε, έχουμε λοιπόν βάση δεδομένων αλλά και δελτία ενημερωτικά τα οποία είναι ευθύνη του, της δικής, του δικού μας τμήματος. Η συνάδελφος Βέρα Μελίσεβιτς τώρα θα σας ενημερώσει και θα σα δώσει κάποια παραδείγματα όσον αφορά τις μελέτες, ιδιαίτερα για την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Από την τελευταία θητεία η Βέρα έχει ε, έχει εμπειρία ελέγχου, λογιστικού ελέγχου. Τότε είναι πολύτιμη για την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Για την προηγούμενη θητεία ε, είχαμε να ασχοληθούμε με διάφορα ζητήματα και με βρία προσέγγιση στον έλεγχο προπολογισμού. Εδώ έχουμε κάποια παραδείγματα που είναι όλα εξαιρετικά. Έχουμε βασίσει την επιλογή στο, κριτήριο αριστείας, διαφοροποίησης και αντικτύπου που είχαν αυτές οι μελέτες, τα εργαστήρια και οι δημοσιεύσεις. Εδώ λοιπόν πρώτη μελέτη ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, ο οποίος ενδιαφερόταν πολύ για αυτό το θέμα και πίεσε ώστε από μελέτη να μετατραπεί σε έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, ώστε να υπάρξει ψήφισμα του, ε, του Ευρωκοινοβουλίου για το πώς χρησιμοποιείται ο ευρωπαϊκός προπολογισμό για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα. Ένα παράδειγμα που μπορεί να σας δείξει πόσο μπορείτε να προχωρήσετε με βάση μια μελέτη τέτοια εάν ε, το επιθυμείτε. Ε, μετά η άλλη μελέτη είναι η αναθεώρηση του κανονισμού Όλαφ. Ε, αυτό το εργαστήριο το προετοιμάσαμε ώστε να προετοιμάσουμε τα μέλη για την αναθεώρηση του κανονισμού της Όλαφ ε, που συμμετείχαν εξαιρετικοί εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί, ε, ποινικού δικαίου, αλλά και εμπειρογνώμονες από την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό το εργαστήριο ε, μετά υπήρχε μια, οδήγησε σε μια μελέτη που αφορά τον Ευρωπαίο Ισαγγελέα και εξετάζει πώς οι δράσεις μη συμμετεχουσών ε, χωρών ή συμμετεχουσών κρατών και πώς η συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών ε, και ε, δικαστικών αρχών μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλά αποτελέσματα. Σας τη συστήνω την ανάγνωση αυτή. Τώρα, το θέμα της απαλλαγής είναι μια ενημέρωση για τους ευρωβουλευτές όπου περιλαμβάνονται τέσσερα σενάρια. Πώς αντιμετωπίσουμε την τρέχουσα κατάσταση και μετά χρησιμοποιήθηκε για τη δουλειά της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού για την απαλλαγή του Συμβουλίου. Είναι ένα έγγραφο το οποίο είναι επίσης ε, ε, χρήσιμο για τη δική σας εργασία. Στην επόμενη διαφάνεια έχουμε κάποιες δημοσιεύσεις ε, που είναι πιο σχετικές ε, λόγω του αντίκτυπου που είχαν στους συναδέλφους στην Επιτροπή. Η πρώτη μελέτη είναι ε, πόσο απόδοση έχει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στην τομέα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Είχαμε λοιπόν και studies από τις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες και διαπιστώσαμε πως χρειάζεται καλύτερη ανάλυση των ε, εκθέσεων διαχείρισης των ευρωπαϊκών αντιπροσωπιών. Το εργαστήριο για την καλύτερη καταπολέμηση της απάτης επίσης οργανώθηκε για να εξετάσει τον αντίκτυπο των εργαστηρίων της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα, καθώς και να εξετάσει τις δράσεις των κατών για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Τελικά, λοιπόν, εντοπίσαμε κάποιες κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των απατών. Τέλος, ενημέρωση για τα κενά και στην ε, βάση δεδομένων ε, TED. Μετά από μια μελέτη όσον αφορά τις διαδικασίες ε, δημοσίων διαχωνισμών είδαμε και συμβάσεις είδαμε πως υπάρχουν προβλήματα στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους δημόσιους διαγωνισμούς και τα κράτη-μέλη ζήτησαν να προχωρήσουμε περισσότερο και να αναλύσουμε το θέμα με περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και να προτείνουμε λύσεις. Η Κομισιόν λοιπόν και οι συνάδελφοι από την DG ε, Περιφερειών ενημερώθηκαν για την ανάγκη ε, βελτιώσεις. Πώς μπορείτε να ζητήσετε λοιπόν αυτές μας τις μελέτες. Ως μονομένα κράτη μπορείτε να προτείνετε προτάσεις στους συντονιστές. Και μετά οι συντονιστές ε, προετοιμάζουν επιστολή ε, για να ζητήσουν ε, τη μελέτη αυτή έρχονται σε εμά στη γενική μας διεύθυνση η προσέγγιση και εμείς ε, στο Τμήμα Πολιτικής ως ε, διοικητική υπάλληλοι ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας, οπότε δηλαδή θα συμμετέχετε στη διαδικασία, θα παρακολουθείτε τη διαδικασία, θα σας ζητήσουμε ε, διευκρινήσεις για να καταλάβουμε ακριβώς τι θέλετε να επιτύχετε και ποιοι, ποιες στοιχεία σας ενδιαφέρουν και θα ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας από την ενδιάμεση έκθεση και την τελική έκθεση για να δώσετε τα σχολεία σας αλλά ε, την ευθύνη για τη διαχείριση αυτού του ε, τη σύμβαση και για την, εφαρμογή, την εκτέλεση της μελέτης, την εκπόνηση της μελέτης. Η πλήρης ευθύνη λοιπόν είναι του Τμήματος Πολιτικής. Θα ήθελα να σας καλέσω να μελετήσετε το κατάλογο μας ε, ε, που έχουμε ετοιμάσει για σας με όλες μας τις δημοσιεύσεις και τις εκδηλώσεις που κάναμε στη διάρκεια της περασμένης θητείας. Θα το βρείτε αυτό εδώ στην είσοδο. Έχετε όλα τα στοιχεία, όλα αυτά είναι ε, επιγραμμικά γνωσιευμένα και μπορείτε να τα μελετήσετε. Ευχαριστώ. Τώρα ο συνάδελφος Αλεσάνδρο Νταλφόνσο που κάθεται εκεί πέρα θα συνεχίσει και θα σας εξηγήσει πώς μπορείτε να ε, έχετε πρόσβαση στα προγράμματα έρευνας και εμπειρογνωμοσύνης ως μεμονωμένα μέλη. Good afternoon. Many thanks uh, for the invitation. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, I will present θα σας παρουσιάσω τρεις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ερευνών στα μέλη. Η Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μάλλον. Η PRS. Πρώτον, μετά από αιτήματα μεμονωμένων βουλευτών, ε, δεύτερον, έχουμε ένα κατάλογο δημοσιευμάτων που καλύπτουν όλους τους τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτον, ε, έχουμε και την πρόσβαση σε πολλές ακόμα πληροφορίες από διάφορες πηγές. Στην υπηρεσία μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε ένα τηλέφωνο για τα μέλη, hotline, που μπορείτε να μας στείλετε τα αιτήματά σας για διάφορες έρευνες που θέλετε, αναλυτικά δελτία, ε, προϊόντα και πληροφορίες και υλικό. Όλα αυτά τα αιτήματα φυσικά τα χειριζόμαστε με εμπιστευτικότητα. Απαντούμε μόνο σε σας για να σας βοηθήσουμε να προετοιμάσετε μια ομιλία, μια συνέντευξη ε, ε, που καλύπτουν όλους τους τομείς πολιτικής. Αυτή η έρευνα μπορεί να δοθεί υπό τη μορφή που εσείς θέλετε και σας βολεύει καλύτερα. Δηλαδή, Γραπτός, αναλυτικά, αλλά και με προσωπικές ε, ενημερώσεις, briefing στα γραφεία σας, ακόμα και τηλεφωνικός. Έχουμε και ένα κατάλογο δημοσιεύσεων που καλύπτουν όλους τους τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα έχουμε 5.000 δημοσιεύσεις και επίκενται και νέες. Γενικά εκδίδουμε κάθε μέρα. Επίσης, μπορείτε να έχετε και alert στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο για να σας έρχονται. Έχουμε διάφορες δημοσίευσεις ε, που καλύπτουν από μεγάλες μελέτες όπως είναι η ετήσια οικονομική και ε, δημοσιονομική επισκόπηση που μπορείτε να δείτε στη διαφάνεια εδώ ή ε, αναλύσεις σε βάθος επίκαιρων θεμάτων όπως είναι ε, ο προπολογισμός βάσει επιδόσεων, performance budgeting, αλλά και ε, έχουμε και δημοσιεύσεις που είναι εσκεμένα πιο ευσύνοπτες αλλά πάρα πολύ ενημερωτικές. Εδώ αριστερά μπορείτε να δείτε ένα σημείωμα που λέγεται at a glance, έτσι, με μια ματιά πριν από κάθε ολομέλεια να έχετε μια ιδέα ε, να ενημερωθείτε για ε, τα μεγάλα ας πούμε χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ή πώς εκτελεί το προπολογισμό. Είναι διάφορε σειρέ αυτέ που έχουμε εκδόσεων και δημοσιευμάτων. Άλλη σειρά είναι η πως εκτελει το προπολογισμο ειναι διαφορες σειρες αυτες που εχουμε εκδοσεων και δημοσιευματων αλλη Αυτά τα briefings, η ενημέρωση γίνεται τακτικά σε φάσεις κλειδιά της νομοθετικής διαδικασίας. Παράδειγμα, αναθεώρηση ε, το, της, ε, του δημοσιονομικού κανονισμού, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ή τα διάφορα προγράμματα, ε, μεταξύ αυτών και τα προγράμματα καταπολέμησης απάτης. αυτή η ενημέρωση, λοιπόν, αυτά τα briefing ενημερώνονται τακτικά. Έχουμε και επίκαιρα θέματα, έτσι, συνόψεις, συμπιλήματα για πρόσφατες δημοσιεύσεις. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε και εδώ στην αίθουσα, στην είσοδο. Βεβαίω, οι δημοσιεύσεις μας δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και με όλες τις φάσεις ε, του κύκλου πολιτικής. Δηλαδή από τη στιγμή που μπαίνει ένα θέμα στην ημερησία διάταξη μέχρι τον τελικό έλεγχο. Και μπορώ να σας δώσω και περισσότερα παραδείγματα. Ευχαριστώ ο συνάδελφος. Ευχαριστώ Αλεσάνδρα. Ε, συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε για την εκλογή σας και εσάς και των αντιπροέδρων. Έχουμε ε, σε τέσσερις φάσεις στη νομοθετική ε, περίοδο. Να σας δώσω μια γεύση των προϊόντων που μπορούμε να σας σερβίρουμε για να γευτείτε κατά τη διάρκεια της θητείας σας αρχίζουμε από την πρώτη φάση, ε, τον ορισμό του θεματολογίου. Ένα καλό παράδειγμα ενός προϊόντος εντός εισαγωγικών που θα σας ενδιαφέρει ως μέλη της Επιτροπής σας είναι ε, η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και το κόστος μη Ευρώπης, ε, όπως λέγεται αυτή η μελέτη. Δηλαδή συγκρίνουμε την κατάσταση τι γίνεται όταν δεν υπάρχει καμία δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι γίνεται όταν υπάρχει δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε τομέα για να συγκρίνουμε την κατάσταση και να δούμε ποια μπορεί να είναι η ευρωπαϊκή υπεραξία. Ε, σε σχέση, ε, δηλαδή είναι ένας αντίστροφος έλεγχος της επικουρικότητας. Ε, η επόμενη φάση, η φάση της διαβούλευσης. This is often the case when there's... Uh, uh, Πολύ συχνά όταν ε, σε κάποιο νομοθέτημα προβλέπεται ενδιάμεση αξιολόγηση ή αναθεώρηση, ε, συχνά μας ζητούν να κάνουμε εμείς μια έκθεση που είναι 8 με 12 σελίδες και να πούμε σε ποιο βαθμό πιστεύουμε ότι η νομοθεσία αυτή ε, ευθυγραμμίζεται με την πραγματικότητα. Γιατί μπορεί ας πούμε να μας έχουν ξεπεράσει οι τεχνολογικές εξελίξεις. Η νομοθεσία είναι κάτι το στατικό, ενώ η οικονομία, ιδιαίτερα η ψηφιακή, είναι δυναμικό. Βλέπουμε γνωμοδοτήσεις διαφόρων ε, φορέων όπως είναι ο επόπτης προστασίας ε, προσωπικών δεδομένων, η Επιτροπή των, των, Περιφερειών συγγνώμη, η ΟΚΕ λοιπά. Λαμβάνουμε υπόψη ε, τις εκθέσεις επίσης και του ελεγκτικού συνεδρίου, ιδιαίτερα τις ειδικέ εκθέσεις για συγκεκριμένα θέματα που μας απασχολούν και με τα οποία, στα οποία εργαζόμαστε ταυτόχρονα. Επίσης βλέπουμε και τι λένε οι ακαδημαϊκές ε, συζητήσεις για αυτά τα θέματα. 8 με 12 σελίδες, ε, πραγματικά μια πολύ καλή βάση και αφετηρία για τους βουλευτές για να ε, συζητούν τα θέματα μεταλόγου γνώσεως όταν φέρνει την πρότασή της κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επόμενη φάση τώρα είναι η νομοθετική αυτή καθ' αυτή. Εκεί εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρότασή της, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για κάποια νομοθετήματα και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό συνοδεύεται από μελέτη σκοπιμότητας. Έχουμε λοιπόν ε, αυτές τις μελέτες εμείς. Στις περισσότερες περιπτώσεις δίνουμε τη γνώμη μας για τη μελέτη αντικτύπου που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καμιά φορά θεωρούμε ότι είναι πολύ καλές, άλλες φορές λιγότερο γιατί εντοπίζουμε κάποιες ελλείψεις ή ε, κάποια θέματα που θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί περισσότερο. Καμιά φορά κάθε τμήμα προετοιμάζει τη μελέτη αντικτύπου, όπως κάναμε με 19 νομικές βάσεις για τα προγράμματα ε, εκτέλεσης του προπολογισμού και δαπανών στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επόμενη φάση είναι η φάση του ελέγχου πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτό για τη δική σας επιτροπή. Αυτό που μπορούμε εκεί να κάνουμε είναι μελέτες εφαρμογής, εκτέλεσης, υλοποίηση. Κοιτάμε τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναλήψεις υποχρεώσεων. Η αντίστοιχη υπηρεσία, το τμήμα στο Συμβούλιο, για να δούμε κατά πόσο αυτές οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν μεταφράζονται σε πραγματικότητα. Και επίσης υπάρχει ένας κατάλογος ε, ευρημάτων του ελεγκτικού συνεδρίου. Στις ειδικές εκθέσεις έχουν ένα checklist και διάφορα θέματα προς εξέταση ε, για την χορήγηση απαλλαγής. Ας πούμε στην απαλλαγή του 2017 τι κάναμε. Είναι γύρω στις 30 αυτές οι ειδικέ εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και εμείς κοιτούμε πώς μπορούμε να τις συνδέσουμε με συζητήσεις σχετικές και θέσεις που λαμβάνει το Κοινοβούλιο. Φυσικά λαμβάνουμε υπόψη και τα δικά σας έγγραφα εργασίας και τις συζητήσεις στις επιμέρους ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές, τα ψηφίσματα της Ολομέλειας και επίσης τις προφορικές και γραπτές ερωτήσεις που υποβάλλουν τα μέλη του Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και τις απαντήσεις της Κομισιόν σε αυτές τις ερωτήσεις. Προσπαθούμε δηλαδή όσο γίνεται να συνδέσουμε τις συζητήσεις του Κοινοβουλίου με τα ευρήματα του ελεγκτικού συνεδρίου και όλα αυτά πάντα στην υπηρεσία της Επιτροπής σας για να έχει νόημα το κεφάλαιο της απαλλαγής στις ειδικέ εκθέσεις, οι εκθέσεις επιδόσεων του Ελεκτικού Συνεδρίου. Τελευταία διαφάνεια. Οι πηγές μας. Έχουμε πάρα πολλές πηγές ε, και ε, υπηρεσίες ενημέρωσης των βουλευτών, πολλές δημοσιεύσεις δικές μας, αλλά ε, έχουμε και συνδρομές σχεδόν ε, σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες, ε, περιοδικά, επιστημονικά έντυπα, databases, ε, βάση δεδομένων κτλ. Έχουμε πάρα πολλά βιβλία και επίσης και μία εφαρμογή για κινητά που δεν αναφέρεται. Μπορείτε στο κινητό σας, στο iPhone, να κατεβάσετε το, τη συγκεκριμένη εφαρμογή και να δείτε τη μελέτη που έχει εκπονηθεί σχετικά. Νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ. Α, ένα τελευταίο που ξέχασα. Αν σας ε, ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες μας, γιατί αυτή ήταν μια πάρα πολύ ε, σύντομη ματιά, μπορείτε να μας βρείτε με το, από το τηλέφωνο, ε, με το mail, ή να μας καλέσετε στο 8800. Νομίζω αυτό το τηλέφωνο ε, έχουμε για να σας βοηθήσουμε και να σας πούμε τι μπορούμε να κάνουμε για σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ρον. Να επαναλάβουμε για χάρη των νέων μελών ότι αν έχετε κάποια ιδέα για κάποιο θέμα όπου η δική σας επιτροπή θα θέλατε να μας ζητήσει κάτι, πολύ ευχαριστώ μιλήστε στον συντονιστή σας και ο συντονιστής μπορεί να το θέσει στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών, όπου βεβαίω όλοι οι συντονιστέ μαζί θα αποφασίσουν. Άρα, μην εγκαταλείπετε τις ιδέες που ενδεχομένως έχετε στη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά αν θέλετε μπορείτε να τις καταθέσετε ήδη πριν να αναχωρήσετε σε διακοπές. Η πρόεδρος Χόλμαϊρ, πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ του, στην ε, Ευρωπαϊκή ε, Κοινοβουλευτική Επιστημονική Υπηρεσία, η οποία μας έχει ήδη προσφέρει πολλές ε, χρήσιμες υπηρεσίες και μελέτες που έχουν στηρίξει την εργασία μας. Ευχαριστώ λοιπόν. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις για την επιστημονική υπηρεσία. Βλέπω ότι όλοι είστε απολύτως ικανοποιημένοι και ικανοποιημένες. Ευχαριστώ και προχωρώ στο επόμενο ε, θέμα, το οποίο είναι το υπαριθμόν 5, ανταλλαγή απόψεων για τις προτεραιότητες της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού για την ένατη αυτή κοινοβουλευτική περίοδο. Η θεμελιώδης, ας πούμε, σκέψη εν προκειμένου, και δεν θα είναι βέβαια η τελευταία αυτή η ανταλλαγή απόψεων, πρόκειται για μια ε, έναρξη των, ε, του προβληματισμού. Έχουμε ακούσει ήδη σήμερα το ελεγκτικό συνέδριο, ακούσαμε εξηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακούσαμε και την δική μας επιστημονική υπηρεσία σχετικά με την συνεργασία που προτείνει. Για μας, ως ε, Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού, σημαντικό είναι να καθορίσουμε προτεραιότητες και να συμφωνήσουμε ποια θα είναι η στρατηγική μας, ποιες θα είναι οι προτεραιότητές μας και οι στόχοι μας. Άρα, μετά από ορισμένε προκαταρκτικές παρατηρήσεις, αντιλαμβάνεστε βεβαίως το βασικό καθήκον μας είναι η απαλλαγή. Συνολικά 53 εκθέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για άλλα θεσμικά όργανα, οργανισμούς ε, και, και ε, κοινοπραξίες. Έχουμε λοιπόν ένα αρκετά ας πούμε φορτωμένο πρόγραμμα έχουμε και τρεις νομοθετικές διαδικασίες στις οποίες συμμετέχουμε το φθινόπωρο. Αφενός την πρόταση για κράτος δικαίου για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μαζί με την Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών. Επίσης ε, την προσαρμογή της νομοθεσίας ε, σε συνεργασία με Όλαφ, κανονισμό Όλαφ και συνεργασία Όλαφ με Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το τρίτο είναι το πρόγραμμα καταπολέμησης τη διαφθοράς στα πλαίσια του ΠΔΠ. Τρει λοιπόν νομοθετικές διαδικασίες. Πέραν αυτών, ε, επιδιώκουμε και συμφωνία με το, ε, Ευρωπαϊκό, με το Συμβούλιο για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Ε, είναι λοιπόν αρκετά πλούσιο το πρόγραμμα για τους επόμενους μήνες. Ε, βέβαια, ε, θα θέσουμε και άλλα θέματα για την εργασία της Επιτροπής μας. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού ήλθε πέμπτη μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ε, συνεδριάσεων. Εμένα η προσωπική μου φιλοδοξία δεν είναι να φτάσουμε στην πρώτη θέση. Αυτό που επιθυμώ είναι να δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τις εργασίες μας. Σήμερα το πρωί έθεσα ας πούμε προσεκτικά την ερώτηση, είπα θέλουμε πραγματικά να ακούσουμε όλους τους γενικούς διευθυντέ ή μας αρκεί να μελετήσουμε τις εκθέσεις τους. Θα θέσω το ερώτημα και στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών, αν πραγματικά δηλαδή θέλουμε να διεξαγάγουμε όλες αυτές ε, τις ακροάσεις και στην πραγματικότητα θα είναι ας πούμε Διαλέξει από καθέδρας που θα κάνουν τα πρόσωπα αυτά, δηλαδή θα έρθουν και θα μας διαβάσουν κάποιες εκθέσει που έχουν ετοιμάσει. Ή μπορούμε να περιοριστούμε στη μελέτη των εκθέσεών τους και να εξοικονομήσουμε τον χρόνο αυτό. Άρα νομίζω οποιασδήποτε ε, προτάσεις εύλογης εξοικονόμηση χρόνου είναι δυνατόν να συζητηθούν. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία επίσης χαρίσαμε πολύ προσοχή, μάλλον προσελκύσαμε την προσοχή με τις διαδικασίες που ακολουθήσαμε και με ορισμένα ταξίδια της Επιτροπής μας, όπως Ελλάδα, Ουγγαρία και Σλοβακία. Και βεβαίως και με τις διαπραγματεύσεις μας για τον Ευρωπαίο Ισαγγελέα. Και ακούστηκε πολύ και το όνομα της Επιτροπής μας. Πολύ χρόνο Αφιερώσαμε επίσης και στην σύνταξη των ειδικών εκθέσεων. Έχω λοιπόν την ερώτηση προς τις και τους συναδέλφους. Βέβαια δεν χρειάζεται σήμερα να ε, ληφθεί ε, τελεσίδικη απόφαση. Έχουμε όμως 45 ειδικέ εκθέσεις. Εάν πρόκειται να γίνει παρουσίαση κάθε μια από τι εκθέσει αυτέ εδώ πλήρω στην Επιτροπή, τότε ασφαλώ θα φτάσουμε πρώτη-πρώτη σε αριθμό συνεδριάσεων. Για το λόγο αυτό, ε, θεωρώ ότι ίσω είναι σωστό να το ξανασκεφτούμε, αν δηλαδή μια ειδική έκθεση, η οποία δεν αναφέρεται ειδικά στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Επομένως δεν άπτεται των θεμελιωδών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας. Τα θέλουμε πραγματικά όλα αυτά τα πράγματα να παρουσιαστούν εδώ ξεχωριστά ή μπορούν να παραμείνουν στις ειδικέ επιτροπές. Σας κάνω κάποιες προτάσεις αν θέλετε να τις σκεφτείτε μέχρι την επόμενη συνάντηση των συντονιστών και να δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε την εργασία μας με τρόπο αποτελεσματικό. Βλέπω σήμερα στα πρόσωπά σας ε, ότι έχουν μείνει οι συνάδελφοι που είναι οι πιο υπομονητικοί και οι πιο επιμελείς. Διότι καμιά φορά είδαμε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία την Ingeborg Γκρέσλε, την πρόεδρο, να κάθεται μόνη της στην αίθουσα. Χωρίς ε, να είναι παρόν κανένας συνάδελφος ή καμία συνάδελφος. Γι' αυτό ε, παρακαλώ και πάλι ε, τις συντονίστες και τους συντονιστές και εδώ ε, στο Προεδρείο, δηλαδή να δούμε πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τον τρόπο εργασίας και είμαι ανοιχτή απέναντι σε οποιαδήποτε πρότασή σας. Θα ήθελα να ακούσουμε τώρα τους συντονιστές, πρώτα τον Ολιβιέ και μετά τον Τόμας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με τα λεγόμενά σας. Νομίζω ότι καλά θα κάναμε να είμαστε λίγο πιο επιλεκτικοί στα όσα εδώ πράττουμε. Εγώ δεν έχω καμία πείρα γιατί είμαι εκλογής ε, βουλευτής και δεν μέλος προφανώς στην Επιτροπή. Αυτό ισχύει και για αυτά που είπατε και εσείς για τις ακροάσεις των Γενικών Διευθυντών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ισχύει επίσης και για τις ειδικέ εκθέσεις που λαμβάνουμε από το ελεγκτικό συνέδριο θα πρέπει να είμαστε σε θέση να βγάζουμε την κεντρική ιδέα ε, για τη δουλειά που εμείς καλούμαστε να κάνουμε στην παρούσα Επιτροπή. Ε, έτσι, να ε, έχουμε ένα τέτοιο επιλεκτικό μηχανισμό για τα όσα θα εξετάζουμε με βάση τα έγγραφα που μας διαβάζονται και τις δυνατότητες για διάφορες ακροάσεις. Δεν θέλω να μπω σήμερα σε λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τις εργασίες της Επιτροπής μας. Νομίζω ότι σιγά σιγά οι νέοι βουλευτές θα πρέπει να συντονίζονται και με τις εργασίες Επιτροπής. Απλώς να αναφέρω κάποιες προτεραιότητες της δικής μας πολιτικής ομάδας, Renew Europe. Θα πρέπει να διαβεβαιωθούμε ε, ότι κάνουμε ένα πολύ ε, σωστό έλεγχο δημοσιονομικό. Έχουν γίνει πρόοδοι ε, και από το ελεγκτικό συνέδριο για τις επιδόσεις, ποιες πολιτικές έχουμε ακολουθήσει, ποιες ήταν οι επιτυχίες, οι αποτυχίες, πώς δαπανούμε τα χρήματα για ποια αποτελέσματα. Αυτή τη μέθοδο θα πρέπει να τη συνεχίσουμε και να συγκεκριμενοποιήσουμε περισσότερο τους δείκτες που χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε πιο ξεκάθαρα όσο γίνεται τι κάνουμε και ε, πού πηγαίνουμε. Το είπε και η Μαρτίνα προηγουμένως, ε, ότι θα πρέπει να μειωθούν οι χρόνοι χορήγησης απαλλαγής ε, ή δυνατόν στο εγγύς μέλλον θα πρέπει να μπορούμε να δίνουμε την απαλλαγή κατά το έτος νη συν ένα. Ε, ας πούμε, ε, αυτό γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Το νησιν 2 είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δυστυχώς ε, αυτή είναι η σημερινή τρέχουσα πρακτική μας. Ε, τρίτη προτεραιότητα, είναι δυνατόν να απλουστεύσουμε τους χρηματοοικονομικούς κανόνες και να βελτιώσουμε τη ευελιξία. όσο πιο περίπλοκοι είναι οι κανόνες, τόσο μεγαλύτερο είναι ο κίνδυνος φάλματος. Έχουμε λοιπόν κάθε συμφέρον να ελέγξουμε ξανά και να επαληθεύσουμε τις διάφορες διαδικασίες. Και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ενδεχομένω να σκεφτούμε να το κάνουμε πενταετές για να συμπίπτει και με το νομοθετικό κύκλο αντί για επταετία. Ε, μας απασχολεί και αυτό. Τέταρτη προτεραιότητα. Θα πρέπει συνεχώς να επιμένουμε στο σεβασμό των θεμελιωδών αξιών κατά την ε, επαλήθευση ε, των ε, οικονομικών δραστηριοτήτων. Θέλω επίσης να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τη γραμματεία μας για τη δουλειά που έχει κάνει, ε, για την μελλοντική μας εργασία κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας που είχαμε πριν τις εκλογές του ζητήσαμε να κάνω αυτή τη μελέτη ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της απάτης αλλά και τον ορισμό της σύγκρουσης συμφερόντων στον δημοσιονομικό κανονισμό. Και επίσης ζητήσαμε να εκπονήσει κάτι και συμφωνούμε όλοι εδώ σε αυτό το, το ανέφερε το πρωί συνάδελφος για τη δική μας συμπεριφορά και στάση που θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο επικοδομητική για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση που έχουμε με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, εδώ και τόσο πολύ καιρό. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία τα είπες. Ευχαριστώ αγαπητή Πρόεδρε. Να μην επαναλάβω όσα είπαν όλοι μέχρι τώρα, γιατί βρίσκω ότι η ατμόσφαιρα είναι ατμόσφαιρα συνεργασίας και χαίρομαι που περάσαμε και κάποιο χρόνο χθες με τους συντονιστές για να μιλήσουμε ε, σχετικά με τη μελλοντική συνεργασία και για τις προτεραιότητές μας και μια συνάδελφό μου σχετικά. Πολύ συχνά μάλιστα το πρόβλημα είναι ότι δαπανούμε χρήματα για κάποιο έργο, παράδειγμα, λιμάνια στην Ισπανία. Θαυμάσιο ε, έργο με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα επιτυχημένο. Κάθε ε, τιμολόγιο ε, ελέγχθηκε και έχει δαπανηθεί σωστά, κανένα πρόβλημα. Όμως η λογική του έργου είναι ότι ταυτόχρονα στέλνουμε χρήματα για να βοηθήσουμε το Μαρόκο να ενισχύσει και αυτό τα λιμάνια του. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι το ε, Μαρόκο μπορεί να προσφέρει πολύ χαμηλότερες τιμές στα καράβια. Επομένως κανένα καράβι δεν θα πάει να πιάσει σε ισπανικό λιμάνι. Όλοι θα πάνε στο Μαρόκο. Μέγα πρόβλημα λοιπόν ότι θα έχουμε ένα νέο ισπανικό λιμάνι με νέα υποδομή αλλά τα χρήματα αυτά τελικά δαπανήθηκαν εις μάτιν. Έχουμε δρόμους που δεν οδηγούν πουθενά. Ξεκινούν από πουθενά και οδηγούν πουθενά. Ε, μεγάλους αυτοκινητοδρόμους. 50-60 χιλιόμετρων. Και δεν βλέπετε αυτοκίνητο να κυκλοφορεί πάνω σε αυτούς. Ή στην Ελλάδα που πήγα εκεί πολλές φορές αποστολές με δίθεν επιτυχημένα έργα. Βλέπετε το μετρό της Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε δαπανίσει πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι γίνεται, λειτουργεί το μετρό. Όλα τα έργα αυτά γίνεται καλή τους ε, διαχείριση. Όχι, εκείνη το πρόβλημα. Η αποτελεσματικότητα λοιπόν. Εάν ζητήσω έκθεση για σφάλματα, ε, για παρατυπίες. Θα δείτε ότι θα είναι μηδενικό το αποτέλεσμα. Δεν θα υπάρχει δηλαδή τέτοιο πράγμα, γιατί κανείς δεν λέει ότι ότι τα χρήματα δεν δαπανήθηκαν ε, σωστά. Και βλέπει κανείς ότι συνεχίζεται κάποια ε, αρχιτεκτονική μελέτη ή δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά η αποτελεσματικότητα των έργων αυτών δεν είναι επαρκής. Και δεν βλέπουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα για πολλά χρόνια. Το άλλο είναι η μεταρρύθμιση της Ένωσης. Οφείλω να ομολογήσω ότι θεωρώ ότι έχουμε πολλούς οργανισμούς. Σε κάθε απαλλαγή συζητούμε πολύ για τους οργανισμούς αυτούς και πώς είναι θαυμάσιες οι επιδόσεις τους και μπράβο τους. Όλοι οι οργανισμοί είναι τέλειοι και έχουμε τους καλύτερους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Αλλά κανένας δεν διαρωτάται ποια είναι η οριζόντια επισκόπηση όλων αυτών των οργανισμών. Βλέπουμε σε πολλές αποστολές στα Ηνωμένα Έθνη, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τους οργανισμούς μάλλον, των ε, Ηνωμένων Εθνών που κάνουν θαυμάσια δουλειά στην Ελλάδα για παράδειγμα. Αλλά γιατί η δική μας ΕΑΣΑ δεν λειτουργεί εκεί, διότι η σύμβαση για τις μεταφραστικές υπηρεσίες τώρα παίρνει τόσο χρόνο, γιατί πολλά πράγματα δεν λειτουργούν και ιδίω η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οργανισμών. Έχουμε πολλούς οργανισμούς που που... στην ίδια πόλη. Αλλά δεν μπορούν να δεν καταφέρουν να συνεργαστούν αποδοτικά μεταξύ τους. οι ε, διευθύνσει προσωπικού μετακινούν κόσμο από τον έναν οργανισμό στον άλλον, αλλά όχι αποτελεσματικά και αποδοτικά. Η απόδοση όλων αυτών θα έπρεπε να είναι σωστός. Όλοι λένε ναι, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για το πώς λειτουργούν ε, το, το, ΣΥΠΟΛ και τα λοιπά, αλλά πώς τελικά λειτουργεί ο Σεντεφόπ, η Europol τον 21ο αιώνα. Χρειάζεται αυτός ο οργανισμός και πώς χρησιμοποιούμε τους πόρους αυτών των οργανισμών. Συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ κρίσιμο θέμα το οποίο πρέπει να λύσουμε σε αυτή την πενταετία και γι' αυτό και εγώ ζητώ μεταρρύθμιση της Ένωσης και έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει καλύτερα να ορίσουμε τη σύγκρουση συμφερόντων. Νομίζω πως έχουμε πολύ πρόβλημα εδώ. Συνεχίζονται οι έρευνες γι' αυτό και είναι απαράδεκτο Πολλοί κόσμος που, που υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει δηλαδή σύγκρουση συμφερόντων να συνεχίζουν να παίρνουν χρήματα από την Ένωση. Ε, ε, δεν, ε, ονόματα δεν λέμε, οικογένειε δεν θίγουμε, αλλά υπάρχει, υπάρχουν προβλήματα και το ξέρετε πολύ καλά. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν στην έρευνα αυτών των υποθέσεων να, παίρνουν, να, να περνά τόσο πολύ χρόνο. Και ε, πολλές αποστολές ε, είχαν εστιάσει σε αυτά τα παραδείγματα. Πρέπει να εστιάσουμε και σε κάποια θετικά αποτελέσματα. Για το μέλλον είναι πολύ σημαντικό ίσως να δούμε κάποια έμπνευση να πάρουμε. Γιατί, ας πούμε, Μπορεί στην Ισπανία κάτι να μην λειτουργεί, ενώ λειτουργεί ας πούμε στη Σουηδία. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί τα χρησιμοποιούν τα χρήματα ας πούμε, στη Φιλανδία με επιτυχία, ενώ σε κάποια άλλη χώρα δεν λειτουργεί. Υπάρχουν επιτυχή προγράμματα, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτών. Κάτι ακόμα που πιστεύω θα πρέπει να δούμε μέσα σε, αυτή, τη θητεία, να βρούμε λύσεις γιατί είναι πραγματικά κρίμα να μην έχουμε την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εδώ και 10 χρόνια. Και πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε στον κόσμο και να λέμε πώς ζητάμε διαφάνεια. Ενώ ένα από τους πιο σημαντικούς θεσμού, οργανισμούς της Ένωσης να μην έχει πάρει την απαλλαγή για 10 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κούς. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Έχω και εγώ να συμπληρώσω μερικά. Ορισμένα επικαλύπτονται με τα προηγούμενα και είναι πάρα πολύ χαρμόσυνο αυτό που συμφωνούμε σε τόσα θέματα. Θα ήθελα να πω κάτι. Με σόκαρε το πρωί που άκουσα ότι δεν υπάρχει απαλλαγή για το Συμβούλιο. Ε, ο προπολογισμό του. Αυτό θα πρέπει να γίνει προτεραιότητα. Να καταφέρουμε κάποια στιγμή να δώσουμε απαλλαγή στο Συμβούλιο. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Ε, με σοκάρει. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, θα πρέπει να σκεφτούμε τι γίνεται με εκείνους τους οργανισμούς που έχουμε, τα agencies, αυτού τους αποκεντρωμένους οργανισμούς που λειτουργούν όντως πολύ καλά και όπου τα τελευταία χρόνια όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει να ελέγξουμε μήπως ευσταθεί νομικά, δεν ξέρω να το κοιτάξει η γραμματεία, αν μπορούμε να κάνουμε εκεί ελέγχους δειγματοληπτικούς. Να μην ελέγχουμε το σύνολο, το 100%, αλλά μόνο ένα τμήμα της διαχείρισης. Εκεί θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η έλεγχη αυτή να μην γίνονται εσκεμμένα, στοχευμένα, αλλά να είναι τυχαίοι οι έλεγχοι αυτοί οι δειγματοληπτικοί και να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες. Ε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να κοιτάζουμε τα διάφορα θέματα και να ελέγχουμε τα διάφορα προβλήματα. Μετά, το τρίτο, θα πρέπει να πω ότι παρακολουθούμε οργανισμούς ε, που κάνουν πολλά πράγματα ε, ίδια με μας που είναι παράλληλα και είναι συνέργεια ε, η δουλειά. Αυτά θα πρέπει να ελέγχονται ας πούμε από καιρό εις καιρό. Και σε ό,τι αφορά το ελεγκτικό συνέδριο δεν μπορούμε εμείς να καθόμαστε και να ελέγχουμε 44 εκθέσεις. Ε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και πάλι θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος δειγματοληπτικού ελέγχου, τυχαίου, για να ε, κοιτάμε. Και ένα τελευταίο που είπε ο κύριος Σαστέλ έχουμε κάποιους κανόνες ε, που είναι πάρα πολύ... Ε, και πάλι σοκαρίστηκα όταν είδα τον τόμο αυτό, που, τον όγκο του δημοσιονομικού κανονισμού. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό μαζί με την Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, για να δούμε και να εξετάσουμε ξανά τους κανόνες και πού μπορούμε να προχωρήσουμε σε απογραφειοκρατικοποίηση, απλούστευση των διαδικασιών και να μην ελέγχουμε το 100% να ελέγχουμε έτσι επιλεκτικά κάποια δειγματοληπτικά όπως σας είπα. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος κανείς ζητεί το λόγο. Όχι. Προς το παρόν. Νομίζω ότι ε, το Σεπτέμβριο θα πρέπει να ασχοληθούμε σε επίπεδο συντονιστών με αυτό το θέμα και να κάνουμε πρόταση στην Επιτροπή μας για να συζητηθεί. Καταρχάς, διαβλέπω ε, το θέμα των δικτών, ότι για την αποτελεσματικότητα των δικτών χρειάζεται συζήτηση, ε, το ζητάτε. Μετά, ε, επιλεκτική έκθεση, μάλλον επιλεκτική εξέταση των ειδικών εκθέσεων, ποιες είναι σημαντικές για μας και ποιες για άλλες επιτροπές επιμέρους. Ας πούμε, το δικαίωμα των επιβατών ε, τα δικαιώματα των επιβατών ε, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία η εκθέση αυτή για τη δική μας Επιτροπή, αλλά για την Επιτροπή Μεταφορών φυσικά ιδιαίτερη. Ε, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε αυτές τις επιμέρους ειδικέ εκθέσεις. Για το Συμβούλιο και την απαλλαγή, νομίζω ότι την τελευταία δεκαετία έχει παγιωθεί ένα καθεστώς. Από πλευράς ε, Συμβουλίου, δεν θέλει να μας δώσει κανία ενημέρωση για τον προϋπολογισμό του, που δεν το θεωρώ και πάρα πολύ σκόπιμο και λογικό, και από την άλλη εμείς ε, ακολουθήσαμε αυτή τη σκληρή γραμμή. Θα πρέπει να το ξαναδούμε το Σεπτέμβριο, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα της απαλλαγής για το Συμβούλιο και ιδιαίτερα. Επειδή και εγώ θα έχω πολλές επαφές με το Συμβούλιο στο εξής, ε, δια της ιδιότητός μου, ε, και με τον αρμόδιο εισηγητή για τον προπολογισμό του Συμβουλίου κάποια στιγμή να δούμε μήπως βρούμε κάποια λύση και για αυτό το θέμα. Δεν απέμπολω την ε, ελπίδα αυτή. Ε, ε, έτσι τα τελευταία χρόνια αυτό έχει βασανίσει πάρα πολύ τη γραμματεία και τα γνωρίζουμε τα θέματα. Για το δημοσιονομικό κανονισμό Έχω ζήσει και δουλέψει για δύο αλλαγέ του δημοσιονομικού κανονισμού και έχω σοκαριστεί και εγώ από τον όγκο αυτό, τον τόμο, το δημοσιονομικό ε, κανονισμό. Και μόνο να το διαβάσει κανείς είναι πάρα πολύ βαρύ, ε, ειδικά όταν δεν είναι κάποιος μοιημένος ή κάποιος γνώστης. Είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακό και καθόλου εύκολο να το κάνουμε. Τώρα θα καταφέρουμε να κάνουμε περικοπές, απλουστεύσεις σε κάτι που έχει παγιωθεί σε 28 κράτη-μέλη τόσα χρόνια. Το έχω ζήσει κάθε φορά. Όλο λέγαμε για πιο αποτελεσματικό, για πιο συνοπτικό δημοσιονομικό κανονισμό και κάθε φορά αυτό διωγγωνόταν. Όπως είναι οι διάφορε νομοθεσίε ελάφρυνση, απογραφειοκτικοποίηση που κάθε φορά προσθέτουν και ένα στρώμα γραφειοκρατίας. Το θέμα είναι τι θέλουμε να κάνουμε, τι σημαίνει για μας αποτελεσματικότητα, τι σημαίνει ουσία και περιεχόμενο, πόσες λεπτομέρειες θέλουμε, σε πόσο βάθος θέλουμε να εξακολουθούμε να εξετάζουμε τα θέματα ή πρέπει να κάνουμε. Υπάρχουν πολλές ε, δυνατότητες και πεδίο για συζήτηση. Είμαι στη διάθεσή σας να συνεργαστούμε στην Επιτροπή προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς άλλο το λόγο. το θα το ξαναπούμε στις 4 Σεπτεμβρίου. Σας βλέπω όλους ανακουφισμένους. Ε, καλές νέες διακοπές, να ξεκουραστείτε και θα το βάλουμε και ως προαπαιτούμενο για το φθινόπωρο καλή επάνωδο, να είστε υγιείς και να ξανάρθετε στις Βρυξέλλες ξεκούραστοι μετά τις διακοπές. Ευχαριστώ πολύ.